αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη, παρακαλώ καθίστε. Καθίστε. Και παρακαλώ λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε σε αυτή τη συνάντησή μας, την διακοινοβουλευτική συνάντηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ευγενικά και ιδιαίτερα θερμά να καλωσορίσω όλους εσάς που είσαστε εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή τη συνάντησή μας, τη διακοινοβουλευτική μας συνάντηση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για να μπορούμε να συμμετέχουμε από κοινού σε μια τέτοια συνεδρίαση εργασίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να να εισαγάγω τη δυναμική και το περιεχόμενο αυτής της διακοινοβουλευτικής μας συνεδρίασης λέγοντας, αναφέροντας δύο λόγια καλωσορίσματος πρώτα και κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις βέβαια. Όλοι γνωρίζετε ότι η 1η Δεκεμβρίου 2009 με την συνθήκη της Λισαβόνας που άρχισε να ισχύει τώρα ισχύει πραγματικά και εφαρμόζεται η συνθήκη της Λισαβόνας. Τερμάτισε, ας το πω έτσι, μια μακρόχρονη συζήτηση, πανευρωπαϊκή μακρόχρονη συζήτηση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη που διεξαγόταν και που διήρκεσε για πάνω κάτω 10 χρόνια περίπου. Αυτή η ολοκλήρωση, αυτή η έκβαση όμως είναι ένα τέρμα είναι η εκκίνηση, το ξεκίνημα ενός απόλυτα καινούριου νέου κεφαλαίου και κατά κάποιο τρόπο επίσης είναι και ένα νέο, τελείως νέο ξεκίνημα για την ευρωπαϊκή διαδικασία και τις διεργασίες με την εισαγωγή και θέσπιση νέων κανόνων του παιχνίδιου. Αυτό σημαίνει ότι σε, μέσα από λιγότερο από ένα χρόνο αυτό, αυτή η συνθήκη της με την Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων άρχισε να ισχύει και εφαρμόζεται πλήρως και οι συνθήκες Λισαβόνας και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχουν σε βάθος και σε μεγάλο βαθμό αλλάξει το νομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτό είναι το όνομα το οποίο καθορίστηκε νομικά και νόμιμα για ένα ολόκληρο πεδίο δράσεων, ένα νέο πεδίο νομοθεσίας και δράσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα. Ένα πράγμα είναι σημαντικό. Για πρώτη φορά είναι απόλυτα σαφές και αναφέρεται ρητά και κάθετα ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα, η ευρωπαϊκή ιδέα, οι ευρωπαϊκές διεργασίες αυτές συνολικά δεν είναι μόνο για την ενιαία εσωτερική αγορά ή το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, ή την... αλλά για την ηθαγένεια, για τους πολίτες που βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι πολίτες βρίσκονται ως άνθρωποι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, με τη δημοκρατική ακριβώς διαδικασία που πρέπει να ενισχύεται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτο και ιδιαίτερα σημαντικό όταν έχουμε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που μετά από την έναρξη σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας απαιτεί ένα νέο πλαίσιο και πλέγμα συνεργασίας, πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παράδειγμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα είναι ο συνομοθέτης στους πιο ευαίσθητους τομείς όπως για παράδειγμα για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στα ποινικά θέματα και στην δίωξη του εγκλήματος. Έχουμε λοιπόν ένα κρίσιμο, σημαντικό, κέριο ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε και διαδραματίζουμε. Αποκινούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, σε όλα τα κράτη-μέλη, στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι ο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 12 τη Συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρω ω παράθεμα. Τα εθνικά κοινοβούλια συνεισφέρουν δραστήρια στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας μέσα στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, στο μηχανισμό αξιολόγησης και στην αξιολόγηση των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 70 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την συμμετοχή και εμπλοκή στην πολιτική εποπτεία της Europol και την αξιολόγηση των δράσεων της Eurojust οι δραστηριότητες αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 85 πάντα της συνθήκης. Και γι' αυτό τον λόγο σε αυτή την διακοινοβουλευτική επιτροπή που συναντάται μέσα στο πλαίσιο των διεργασιών που ξεκίνησαν, ξεκίνησαν από τις, ε, τους αρχηγούς, ε, τους επικεφαλής των εκνοβουλίων που συνήθαν στη Στοκχόλμη το Μάιο του 2010. Αυτά όλα μας υπενθυμίζουν τη σημασία, τη σπουδαιότητα της ε, συγκυρίας και της ευκαιρίας αυτής που προσφέρεται ώστε οι πρόεδροι των κοινοβουλίων των κρατών μελών να έχουν ζητήσει από την Βελγική Προεδρία να εξετάσει περαιτέρω την πρόταση για να διεξάγονται σε τακτά διαστήματα οι συνεδριάσεις ε, όσον αφορά τις ε, εσωτερικές υποθέσεις και υποθέσεις δικαιοσύνης, ε, εξωτερικές υποθέσεις. Το Βελγικό Κοινοβούλιο θα υποβάλει τις προτάσεις του στην επόμενη σύνοδο των Προέδρων των Κοινοβουλίων που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2011. Αυτό είναι το πλαίσιο και η συγκυρία, ο ιστός εντός εισαγωγικών αυτής της συνεδρίασής μας. Αυτή η συνεδρίαση είναι ακριβώς μια συνεισφορά όσον αφορά την εντολή που δόθηκε από τους Προέδρους των Κοινοβουλίων και από το Βελγικό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Λίμπε Committee και ως αρμόδιος για τέτοια ευαίσθητα θέματα που συσχετίζονται με το χώρο ελευθερίας, ε, δικαιοσύνης και ασφάλειας, απόλυτα κατανοώ τις ευθύνες ε, που έχουμε ενώπιον των πολιτών μας και ενώπιον όλων των άλλων ατόμων που προστατεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι μεγάλη πρόκληση να νομοθετεί κανεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερία και της ασφάλειας. Μια και πρέπει ταυτόχρονα πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τις βέλτιστες πιθανές λύσεις, δυνατές λύσεις, διασφαλίζοντα και διατηρώντα όμω τα στοιχεία των εθνικών νομικών τάξεων και πλαισίων. Πουθενά αλλού δεν είναι τόσο σημαντικό η αρχή επικουρικότητας και η αρχή της αναλογικότητας να γίνονται απόλυτα σεβαστές με την πλήρη συμμετοχή των εθνικών νομοθετών από πλευρά των κοινοβουλίων. Αυτό αληθεύει επίσης και για τις λειτουργικές πτυχές, για την λειτουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο και συγκυριακό ότι πρόσφατα αρκετές ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα όπως το SIS, Schengen Information System, το σύστημα πληροφοριών Schengen και η Eurodac όσον αφορά το Visa Information System, VIS, το σύστημα θεωρήσεων διαβατηρίων. Δημιουργήθηκαν όλα αυτά ως κοινά εργαλεία, σε ένα κοινό χώρο, για να μπορούμε να λειτουργούμε και να ερχόμαστε σε επαφή και να δρούμε μεταξύ των κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υιοθετώντα αυτές τις συστάσεις το 2009 για το πρόγραμμα της Στοχόλμης, κατέστησε σαφές τον κατεπήγοντα χαρακτήρα της ενίσχυσης της δημοκρατίας, δημοκρατικότητας λογοδοσία και υπευθυνότητα όσον αφορά τον χώρο της ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μέχρι το Σεπτέμβριο 2010 τις νέες νομοθετικές προτάσεις που θα αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας για την Europol, την Eurojust και την συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια γενική αξιολόγηση όλων αυτών των πτυχών για τον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Μετά από ένα χρόνο από την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμη υλοποιήσει αυτή την υποχρέωσή της, αυτό το αίτημα ή την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν την έχει υλοποιήσει ακόμη. Ξεκινήσαμε όμως παρόλα αυτά τις συζητήσεις κοινοβουλευτικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις για την μεταρρύθμιση του ε, πλαισίου λειτουργίας της ε, Europol, της Ευρωπόλ. Για αυτούς όλους τους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει προγραμματίζει τις νομοθετικές της, προτα... νομοθετικές της προτάσεις πριν από το 2013. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι η σημερινή νομική, νομοθετική κατάσταση που αναφέρεται στη συνθήκη της Νίκαιας Μέχρι τότε ουσιαστικά θα μπορέσει να επιβιώσει. Αν υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια πρόταση το 2013, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας ως Ευρωκοινοβούλιο να ολοκληρώσουμε όλες τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ένα έτος. Και έτσι διακυβεύουμε να χάσουμε την πενταετή περίοδο που καθορίζεται από το πρωτόκολλο 36 για την λησβονοποίηση θα έλεγα, για την ε, ευθυγράμμιση με τις αρχές της συνθήκης Λισαβόνας. Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Είμαστε όλοι πεισμένοι ότι ακόμα και αν είναι εύλογο να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πρόσφατες αποφάσεις για τη Europol και τη Eurojust λειτουργούν και θα πρέπει μέχρι τα μέσα του 2011 να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες και μετέπειτα θα πρέπει να ξεκινήσει το νομοθετικό έργο από πλευράς μας. Στο μεσοδιάστημα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν ισχύει, διότι ισχύει φυσικά ισχύει και είναι λειτουργική η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει να επιτύχουμε όμως κάποιες πραγματιστικές, ρεαλιστικές λύσεις που θα καταστήσουν εφικτό και δυνατό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα άτυπο πλαίσιο όπου οι εθνικοί εκπρόσωποι, οι συγητέ και σκιώδεις οι της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα μπορούν να δρουν ελεύθερα και να έχουν σχέσεις και επαφές και διαβουλεύσεις με τους ομολόγους τους όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Και αυτή η λογική, αυτό το πρότυπο θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τους οργανισμούς και τις τα κέντρα και τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται όπως ε, το Γραφείο Υποστήριξης ε, Ασύλου ΕΣΟ και η Frontex για παράδειγμα υπηρεσία φύλαξη εξωτερικών συνόρων. Και τέλο, εξίσου σημαντικό, τα εθνικά κοινοβουλία θα πρέπει να παρακολουθούν όλε αυτέ τι δραστηριότητε. Αυτό τι σημαίνει. Παρακολούθηση των δικτύων όσον αφορά και την ανταλλαγή πληροφοριών που θα μοιράζονται τα κράτη-μέλη, τρίτε χώρε και διεθνεί οργανισμοί και ε, φορείς. Για αυτούς όλους τους λόγους αποφασίσαμε να εισαγάγουμε τα κυριότερα σημεία στο σεμινάριό μα, το, Schengen, το σύστημα Schengen που είναι το πιο ισχυρό εργαλείο και μέσο για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με όλες αυτές τις παρατηρήσεις λαμβανομένων όλων αυτών υπόψη και γνωρίζοντας ότι μόλις ξεκινήσαμε όλη αυτή την, αυτό το έργο και το εγχείρημα έχουμε μια δυναμική που πρέπει να διατηρηθεί και να τροφοδοτείται για αυτή την πενταετή περίοδο που έχουμε μπροστά μας ενώπιόν μας να εγγράψουμε λοιπόν για αυτή την περίοδο στις ατζέντε μας, στις, ε, στα, ημερολόγιο μας στα ημερολόγιο μας, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε όσον αφορά και τον τρίτο πυλώνα, όσον αφορά τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς που συσχετίζονται με τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Και πρέπει, πρέπει εδώ να δηλώσω και να πω ρητά ότι Είμαστε ικανοποιημένοι, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι συναντώμεθα σε αυτά τα κτίρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους εκπροσώπους των 27 εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον 18 κράτη-μέλη που είναι παρόντα σήμερα εδώ, εκπρόσωποι 18 κρατών μελών που είναι σήμερα εδώ παρόντες. Για να προχωρήσουμε θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κούκελμπεργκ πρώτα από πλευράς του Συμβουλίου που θα παρουσιάσει τις θέσεις του Συμβουλίου και μετά, μετά την δική του παρέμβαση, την εισήγησή του θα δώσω τον λόγο στη συνέχεια στον κύριο Μπρόβερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κούκελμπεργκ έχετε τον λόγο λοιπόν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συστηθώ να ολοκληρώσω δηλαδή την παρουσίαση που μου έκανε ο Πρόεδρος. Είμαι ο Ασκόν την Προεδρία κατά την Βελγική Προεδρία ε, του ΚΟΖΙ της Μόνιμης Επιτροπής ε, Λειτουργικής Συνεργασίας για θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη ΛΥΜΠΕ και πιο συγκεκριμένα τον Πρόεδρο, τον κύριο, τον ε, κύριο Λόπες που με κάλεσε Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές αλλά και τους Εθνικούς ε, Βουλευτές για την παρουσία τους ε, εδώ σήμερα όπως επίσης και για το ενδιαφέρον το οποίο παίρνουν για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο μου τιμή μου αλλά και καθήκον μου ως προεδρεύον του ΚΟΖΗ να έρθω εδώ να αναφέρω στα Εθνικά Κοινοβούλια για τις ε, εργασίες της ε, Λειτουργικής Επιτροπής. Λοιπόν, είναι τιμή και θα σας το πω γιατί, αλλά και υποχρέωση, διότι η μέσω της ε, δράσης της θα πρέπει να έχει μια θετική επίπτωση στην ασφάλεια, αλλά και στην ελευθερία και στην ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια απόλυτη διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου. Όπως ε, μου ζήτησε η Επιτροπή Λιμπέ να σας ε, αναφέρω σε τι, τι ρόλο παίζει το ΚΟΖΙ για την ε, συνεργασία των ευρωπαϊκών οργανισμών. Να σας παρουσιάσω λοιπόν το κόζι αυτό κάθε αυτό, τις βάσεις του, τις αρμοδιότητες του, τις αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να βασίζεται ε, το κόζι για να μπορέσουμε να περιχαρακώσουμε τις αρμοδιότητές του γιατί το όργανο είναι απόλυτα καινούριο. Θα σας αναφέρω επίσης και το πρόγραμμα του κόζι μέχρι τα τέλη του τρίου δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011 και πέρα βέβαια από αυτή την ημερομηνία διότι οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι στόχοι που ξεπερνούν την Βελγική Προεδρία και ίσως και την Ουγγρική Προεδρία. Θα ξεκινήσω λοιπόν παρουσιάζοντας το κοζί. Να σας θυμίσω την νομική βάση που αποτελεί δηλαδή και την βασική γραμμή λογικής που κράτησε η Βελγική Προεδρία για να ορίσει τις ε, θέσεις της και κατά τη Βελγική Προεδρία αλλά και να προετοιμάσει την Ουγγρική Προεδρία. Πρώτον, το άρθρο 71 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι το ΚΟΖΙ δημιουργείται για να διασφαλίσει μέσα στην Ένωση την πρόθεση και, και την ενίσχυση της ε, λειτουργικής συνεργασίας για εσωτερική ασφάλεια. Μετά έχετε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης το οποίο είναι θεμελιώδες έγγραφο για θέματα συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. και όπου θεωρεί ότι θα έπρεπε να καταστεί η εσωτερική ασφάλεια μία από τις πρώτες βάσεις του ΚΟΖΗ. Και μετά έχουμε και μία απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου του 2010, είναι πάρα πολύ πρόσφατη, που <coughs> δημιουργεί το ΚΟΖΗ και ορίζει και την γενική του αποστολή. Δηλαδή, μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται Συμβούλιο, Οργανισμοί, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. Να σας πω τώρα μερικά πράγματα. Άρθρο 2. Ενισχύει και προωθεί τον συντονισμό των λειτουργικών δράσεων των κρατών μελών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Ε, αυτός είναι ο γενικός ορισμός. Πρόκειται όμως ε, για μία πολύπλευρη ε, αρμοδιότητα και υπάρχει και μία μεγάλη ποικιλία ενδιαφερόντων, διότι εμείς εδώ μιλάμε για εσωτερική ασφάλεια, σε γενικό επίπεδο μιλάμε για δικαστικά θέματα, μιλάμε για αστυνομικά θέματα, αλλά μιλάμε όμως και για πολιτική άμυνα, για ασφάλεια των συνόρων. Υπάρχουν λοιπόν πολλές προβληματικές μέσα σε αυτήν την Επιτροπή Λειτουργικής Συνεργασίας. Άρθρο 3 λέει ότι το ΚΟΖΙ διασφαλίζει συνεργασία και λειτουργικό, πραγματικό λειτουργικό συντονισμό στα πλαίσια του άρθρου 5 του τμήματος 3 της συνθήκης. Συνεχίζει το άρθρο 3. Αξιολογεί το ΚΟΖΙ το γενικό προσανατολισμό και την αποτελεσματικότητα της λειτουργικής συνεργασίας. Διαπιστώνει ποια είναι τα κενά και οι λήψεις του συστήματος και αν υπάρχουν προβλήματα τότε το αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές για να τα διορθώνει. Το κόζι ε, βοηθάει το Συμβούλιο σε όλα τα θέματα που αφορούν στη ρήτρα αλληλεγγύης. Δεν συμμετέχει στις επιχειρήσεις. Εγώ μιλάω για λειτουργικότητα, αλλά δεν έχουμε... Ε, δεν είμαστε αυτοί που συμμετέχουμε. Μπορούμε ίσως να συντονίσουμε, αλλά δεν συμμετέχουμε. Επίσης το ΚΟΖΙ δεν συμμετέχει στην επεξεργασία νομικών πράξεων. Τις νομικές πράξεις τις επεξεργάζονται άλλα όργανα, όχι το ΚΟΖΙ. Το ΚΟΖΙ είναι ένα λειτουργικό όργανο. Άρθρο 5 είναι πολύ σημαντικό για το θέμα που μας αφορά γιατί λέει ότι εκπρόσωποι της Eurojust, της Europol, του Frontex και άλλων αρμοδίων οργανισμών καλούνται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του ΚΟΖΗ. Και λέει ότι το ΚΟΖΗ θα, θα συμβάλλει στην συνοχή της δράσης αυτών των οργανισμών. Δηλαδή είμαστε εδώ για να παίξουμε και έναν συντονιστικό ρόλο, για να πετύχουμε το optimum από αυτούς τους οργανισμούς. Έχουμε εδώ την απόφαση της 25ης Φεβρουαρίου, αλλά μπορεί να προκύψουν και άλλες με τα άρθρο 6. Το ΚΟΖΙ υποβάλλει τακτικά στο Συμβούλιο μια έκθεση για τις δραστηριότητές του και στο τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πληροφορούνται από το Συμβούλιο για τις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής. Αυτό εξηγεί δηλαδή και για ποιο λόγο βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και το ξαναλέω τιμή μου και χαρά μου. Πιο πολύ από ό,τι καθήκον. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα στο πρόγραμμα εργασίας που υπέβαλε η Βελγική Προεδρία στα μέλη του ΚΟΖΗ στις 25 Ιουνίου του 2010 και το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου. Και αυτό πολύ πρόσφατο λοιπόν. Αυτό το πρόγραμμα το επεξεργαστήκαμε βάσει των τριών κειμένων που αναφέρομαι, είπαμε, σε συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία, για να είμαστε σίγουροι δηλαδή ότι θα υπάρχει μία συνέχεια σε αυτά τα οποία θα προτείνουμε και θα πράξουμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολυετές, το οποίο δεν δεσμεύει μόνο την Βελγική και την Ουγγρική Προεδρία, αλλά και τις επόμενες Προεδρίες. Αυτό το πρόγραμμα το ζήτησαν πολλές αντιπροσωπείες, από τότε δηλαδή που συγκροτήθηκε το ΚΟΖΙ από την πρώτη του συνεδρίαση το Μάρτιο φέτος. Εγώ πιστεύω ότι εκπληρώσαμε πολλές επιθυμίες όταν ε, ε, προχωρήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, λάβαμε υπόψη μας μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, βασικές αρχές. Ε, διδαχτήκαμε από το παρελθόν, από τις εργασίες προετοιμασίας της Λισαβόνας. Και φυσικά εμπλουτίζουμε, εμπλουτίζουμε τις αρχές μας και από την εμπειρία των συνεδριάσεών μας μια φορά το μήνα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε συνέπεια συνέχεια, διότι εμπνεόμαστε από αυτά που είχε ετοιμάσει η Ισπανική Προεδρία. Προστιθέμενη αξία. Τα θέματα συζητιούνται στο κόζι, αν το κόζι είναι σίγουρο ότι μπορεί να προσφέρει κάτι, να γνωμοδοτήσει, να δώσει συστάσεις και είναι θέματα που δεν έχουν συζητηθεί σε άλλη ομάδα Λοιπόν, ολιστική θέση. Σας ανέφερα λοιπόν τις, ε, ε, τα διάφορα θέματα που απασχολούν το ΚΟΖΙ και όταν συζητάμε για ένα θέμα εσωτερικής ασφάλειας λαμβάνουμε υπόψη όλους τους ενδιαφερόμενους και όλα τα ζητήματα που συνδέονται σχετικά. Ούτως ώστε λοιπόν όλοι να αποτελούν μία αλυσίδα. Επίσης θέλουμε να είναι ρεαλιστικοί και συγκεκριμένοι η θέση μας με αυτά αποτελέσματα. Αυτό το λέω τακτικά σε πολλά διεθνή φόρουμ. Είναι θέμα δηλαδή αξιοπιστίας όλων αυτών των φόρουμ να καταλήγουν πάντα σε κάτι συγκεκριμένο όμως. Θέλουμε λοιπόν εμείς στο τέλος των εργασιών μας να αποδείξουμε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς που σας απαρίθμησα πριν αλλά και στους πολίτες της Ένωσης ότι κάτι κάναμε. Και στο τέλος ε, φυσικό θέλουμε να έχουμε και μία επίπτωση στην ευρωπαϊκή εσωτερική ασφάλεια. Για να επεξεργαστούμε λοιπόν το πρόγραμμά μας συνεργαστήκαμε με συνεργασίες και διαβουλευθήκαμε με όλους γύρω από το τραπέζι του Κόζη και με τρόπο διαφανή. Εμείς ε, σεβόμενοι τη συνέχεια λάβαμε υπόψη μας το τι πραγματοποιήθηκε από την Ισπανική Προεδρία και μετά καλέσαμε και όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, την Κομισιόν, τους οργανισμούς για να μας υποβάλουν προτάσεις θεματικές ε, προτάσεις οι οποίες θα είχαν και μια λειτουργική ε, πρόπτικη και θα μπορούσαν να δώσουν μια προστιθέμενη αξία. Λάβαμε λοιπόν 34 ε, προτάσεις από τα κράτη-μέλη, από τη γραμματεία από την Κομισιόν, από το Γενικό Γραμματέα κτλ. Εμείς τις ξεδιαλέξαμε αυτές τις 34 προτάσεις και καταλήξαμε σε ένα μικρότερο κατάλογο 14 βασικών θεματικών. Είναι μικρός ο κατάλογος ως προς τον αριθμό των θεματικών, θα σας αναφέρω όμως μερικά από αυτά τα θέματα που είναι πολύ φιλόδοξα. Εμείς δεν θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε 50-60 διαφορετικά θέματα, γιατί γιατί θελήσαμε να μην μείνουμε με άδεια τα χέρια στο τέλος αν ξεδιαλέγαμε πολλές προβληματικές. Λοιπόν, πρώτος στόχος μας από αυτούς τους 14 είναι ο συντονισμός των διαφόρων οργανισμών. Δεύτερο, ένα ευρωπαϊκό policy cycle, ένα δηλαδή, ένας πολιτικός κύκλος. Δεν ξέρω πώς θα το έλεγα στα γαλλικά το policy cycle. Μιλάμε για το σχέδιο αρμονία μέσα με τη δικιά μας ορολογία. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προωθεί σε αυτό το εξάμεινο η Βελγική Προεδρία και έχει ως στόχο να αναπτύξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία σταθερή και επιστημονική και στεναρή μέθοδο εργασίας που να λαμβάνει υπόψη όλες τις απειλές προς την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης και που θα επιτρέπει στους υπουργούς όταν αυτοί θα πρέπει να ορίζουν τις προτεραιότητες της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης να βασίζονται σε μία μέθοδο η οποία θα είναι δοκιμασμένη και θα τους επιτρέπει να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους. Θα επιτρέπει λοιπόν να διαμορφώνουμε εμείς αυτή τη λίστα που θα δίνουμε στους υπουργούς και που θα διαμορφώνουν τις στρατηγικές τους. Δεν θέλουμε ένα νέο μέσο, θέλουμε να τακτοποιήσουμε, να συντονίσουμε και να εναρμονίσουμε τα διάφορα μέσα προβλέποντας κιόλας λίγο πολύ τα ρίσκα εμείς μιλήσαμε ότι καταρχήν θα έπρεπε να ορίσουμε την, ε, το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, τι μορφές παίρνει αυτό το έγκλημα και πώς θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε στους επόμενους μήνες. Ένα τρίτο παράδειγμα, η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας που όπως σας το έλεγα και μέσα στα πλαίσια της Στοκχόλμης αποτελεί κεντρικό πυρήνα των ανησυχιών του Κόζη. Συνεργαστήκαμε με την Κομισιόν σχετικά, η οποία θα πρέπει να κάνει μια σχετική ανακοίνωση το Νοέμβριο νομίζω. Το κόζι θα βασιστεί λοιπόν στην ανακοίνωση της Κομισιόν και θα προχωρήσει στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση αυτής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Αύριο 5 Οκτωβρίου συνεδριάζει στο Κόζι και το απόγευμα αύριο θα έχουμε και μία συζήτηση με την Κομισιόν για το σχέδιο επικοινωνίας. Ανυπομονώ λοιπόν να έρθει αύριο το απόγευμα. Τέταρτο παράδειγμα είναι η καταπολέμηση κατά του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών στο Κόζι συμφώνησαν και είπαν ότι η εγκληματικότητα μας απασχολούσε όλους, το οργανωμένο έγκλημα μας απασχολούσε όλους. Και είπαν όλοι να κάτσουν να το σκεφτούν, να προβληματιστούν. Δηλαδή για να δούνε ποιοι είναι οι μηχανισμοί καταπολέμησης και πρόληψης αυτής της εγκληματικότητας. Και όχι μόνο δηλαδή την ποινική κατασταλτική πλευρά δεν θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε εμεί μόνο τις ποινικέ κυρώσεις, αλλά να δούμε και εναλλακτικού ε, ε, τρόπους όπου ας πούμε το ε, διοικητικό δίκαιο που επιτρέπει την κατάσχεση αγαθών, που επιτρέπει το κλείσιμο ε, ορισμένων οργανισμών Τέλο πάντων αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε με την ε, Ουγγρική Προεδρία και αποτελεί και μια προτεραιότητα δηλαδή τη Ουγγρική Προεδρία. Πάμε τώρα στον συντονισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών. Ποιο είναι ο ρόλος του ΚΟΣΥ για τα θέματα συντονισμού. Είναι το άρθρο 5 της απόφασης του Συμβουλίου τη 25 Φεβρουαρίου του 2010 που επιτρέπει στο ΚΟΖΙ να διασφαλίζει τη συνοχή της δράσης αυτών των οργανισμών. Πρόκειται λοιπόν για ένα συντονιστικό ρόλο, ούτως ώστε αυτές οι εργασίες, αυτοί οι οργανισμοί να εργάζονται με τον εξαιρετικότερο τρόπο και στην πρώτη συνεδρίαση της 11ης ε, Μαρτίου το είχαμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη και συζητήθηκε το θέμα και στις 30 Τετάρτου και στις 25 Ιουνίου. Εμείς θεωρήσαμε λοιπόν το συντονισμό των ε, οργανισμών ως ένα από τα θεμελιώδη σημεία της Βελγικής και Ουγγρικής Προεδρίας. Οι οργανισμοί που γνωρίζουμε, τουλάχιστον αυτούς που θα δείτε εδώ πέρα, Όλες έχουν μια συγκεκριμένη εντολή με διαφορετικές ευθύνες και στόχους. Αλλά καμία από αυτές μόνη της δεν μπορεί να αναπτύξει μόνη της την όλη της δυναμική χωρίς τη βοήθεια των άλλων οργανισμών και την ενίσχυση των κρατών μελών. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς λειτουργούν, πώς συνεργάζονται και αυτό σεβόμενοι και τις αρμοδιότητες των άλλων υπηρεσιών της ε, Ένωσης και έχω κατά νου εδώ και την Κομισιόν. Αλλά ο εξεξιών ε, συνάδελφος θα τα πει μετά αυτά. Για το συντονισμό λοιπόν ε, των, ε, των οργανισμών αποφάσισε το Τζάι την 1η Οκτωβρίου του 2009 όταν η Σουηδική Προεδρία ζήτησε από την Ευρωπόλ, την Eurojust, το Frontex και τη ΣΕΠΟΛΑ να ετοιμάσουν κατευθυντήριε γραμμές για τη στρατηγική και λειτουργική εργασία, να ορίσουμε κοινέ προδιαγραφές, να, πάρουμε, να αναλάβουμε κοινέ πρωτοβουλίες για θέματα κατάρτισης, να αναπτύξουμε τις μεθόδους εργασίας και τον τρέχοντα τρόπο δουλειάς για να έχουμε στην πράξη συνεργασία. Καταφέραμε λοιπόν να έχουμε μία κοινή έκθεση στα τέλη του 2009, αρχές 2010. Είναι η πρώτη φορά που οι τέσσερις οργανισμοί παρουσιάζουν ταυτόχρονα μία έκθεση, μία κοινή έκθεση για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Έχουμε μία προσωρινή έκθεση που υποβλήθηκε στο ΚΟΖΗ στις 11 Μαρτίου του 2010, δηλαδή στην πρώτη συνεδρίαση. Και διαπιστώσαμε ε, ότι υπήρχε μία καλή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, αλλά κυρίως διμε, διμερός. Ε, επίσης, φαινόταν από αυτή την έκθεση ότι χρειάζεται ένας ορθολογισμός ε, της δράσης Λοιπόν, στις αρχές ε, Απριλίου είχαμε την τελική έκθεση και αναφέρονται τα υπάρχοντα πρωτόκολλα και συμφωνίες σε διμερές επίπεδο, εξαγγέλλονται διάφοροι στόχοι για να βελτιωθούν αυτά τα πρωτόκολλα και ορίζονται και τομείς ε, για τους οποίους θα μπορούσαμε να συνάψουμε νέους συμφωνίες. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκεκριμένα και πολυμερός. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το συγκεκριμένο, κάτι το πρακτικό. Πρόκειται για ένα κείμενο ιδιαίτερα ευανάγνωστο με συγκεκριμένους στόχους. Είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο κείμενο. Δεύτερον, αυτή η έκθεση λαμβάνει απόλυτα υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Και τρίτον, αναφέρεται σε προβληματικές που οι οργανισμοί μπορούν να λύσουν μόνοι τους. Κάνανε μία αυτοανάλυση και αυτοακριτική. Ανέσυραν νέους στόχους, νέες προκλήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά πρόκειται για στόχους που μπορούν να υλοποιήσουν μόνοι τους αυτοί οι οργανισμοί. Επίσης, επίπεδο δεν αποκλείεται αυτού του είδους οι δράσεις να διευρυνθούν και σε άλλους οργανισμούς που αφορούν στην εσωτερική ασφάλεια, ας πούμε ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαίωμα, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο ή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικής Κατάρτισης. Τώρα, ε, είδατε, ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν και άλλους οργανισμούς ως παρατηρητές. Τώρα, για την διμερή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις λειτουργικού χαρακτήρα ανταλλαγή πληροφοριών, ανάλυση, αξιολόγηση της απειλής, κοινέ ανακριτικές ε, επιτροπές, κατάρτιση, εξωτερική επικοινωνία. Και οι οργανισμοί που θα μιλήσουν σε λίγο μπορούν να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, πολυμερείς συμφωνίες να έχουν πιο στρατηγικό χαρακτήρα και θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στην καθημερινή συνεργασία και στη λειτουργία, αλλά μακροπρόθεσμα συνολικά στην εσωτερική ασφάλεια. Να σας αναφέρω μερικούς από αυτούς τους στόχους να αναπτυχθούν μέτρα που θα επιτρέπουν να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή, συνέχεια διαλειτουργικότητα μεταξύ των οργανισμών, να δημιουργηθεί μια κοινή σφαίρα διαχείρισης με συνεδριάσεις μεταξύ ε, ηθινόντων, κοινή προσέγγιση για τα θεσμικά ευρωπαϊκά ζητήματα και τις εξωτερικές σχέσεις, ε, συνδυασμός προσπαθειών στην έρευνα και στην ανάπτυξη, κοινέ προσπάθειες στον τομέα της κατάρτισης δημοσιοποίηση των εργασιών ε, των οργανισμών. διότι υπάρχει μία σαφής άγνοια για το πώς λειτουργούν οι διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα τονίζουμε. Τελευταίο, να αποδειχθεί, ε, συγγνώμη, να ενισχυθεί η διαοργανική συνεργασία μέσα από συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και ε, δράσεις πληροφόρησης. Αυτοί είναι οι στόχοι που θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη συνέργεια, να μην έχουμε επικαλύψεις και να μπορούμε να έχουμε μια optimum χρήση και αξιοποίηση των οργανισμών. Τώρα για τα θέματα επικαιρότητα του ΚΟΖΙ σχετικά με αυτούς τους οργανισμούς. Λοιπόν, μετά από την τελική παρουσίαση της έκθεσης των οργανισμών, το ΚΟΖΗ αποφάσισε στις 25 Ιουνίου να καλέσει τους οργανισμούς να εφαρμόσουν τα περισσότερα από τα μέτρα που ανέφερα στην τελική έκθεση, να διαμορφώσουν μια κοινή σφαίρα συναντήσεων μεταξύ των ηθινών των και θα προεδρεύονται αυτές οι συνεδριάσεις από τον διευθυντή του οργανισμού που υποδέχεται τη συνεδρίαση. Όπως επίσης θα συμμετέχουν και αρμόδιοι από τους άλλους οργανισμούς. Και τα πρακτικά βεβαίως θα έρχονται στο ΚΟΖΗ. Πρώτη συνεδρίαση στις 26 Ενδεκάτου στη Χάγη που θα συμμετέχουν αυτοί που σας ανέφερα και εγώ θα συμμετέχω. Και ολοκληρώνω. Θα διαπιστώσατε τι σημασία δίνει το ΚΟΖΗ στην, στο συντονισμό της συνεργασίας των οργανισμών. Θα το σπρώξουμε ούτως ώστε να προχωρήσουμε, η Βελγική Προεδρία δηλαδή, να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Κούκελμπεργκ. ο οποίος εκπροσωπεί τη Βελγική Προεδρία αλλά είναι και πρόεδρος του ΚΟΣΥ. Σας ευχαριστώ πολύ αν μας στείλετε την κοινή έκθεση την οποία αναφέρατε, δηλαδή της Europol, της ΕΠΟΛ, του Frontex κλπ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ντεμπρεβέρ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω, βλέποντας το ρολόι μου, ότι θα μιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να είμαι σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ θα ήθελα στην αρχή αυτής της σύντομης παρουσίασης να σας ε, κάνω τρεις υπομνήσεις που θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Πρέπει να τις έχετε κατά νου αυτές τις δύο ημέρες εργασιών και αποφάσεων. Θα συζητήσετε εθνικά κοινοβούλια και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα ένας διαθεσμικός διάλογος γίνεται ταυτόχρονα σχετικά με το ρόλο, την αποστολή και τον έλεγχο των οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο διαθεσμικός διάλογος ζητήθηκε μετά από μία ανακοίνωση της Επιτροπής του 2008. Δεδομένου ότι είναι και διαθεσμικός ο διάλογος, εισπυρώνει Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν. Θα καταλήξει σίγουρα το 2011 σε συμπεράσματα είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε μία συγχρονία και συντονισμό αυτών των δύο πραγμάτων, δηλαδή του διαθεσμικού διαλόγου και, των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης. Και να σας θυμίσω και τι είπε ο κύριος Κούκελμπεργκ. Πρέπει να είναι καθαρό στο κεφάλι του καθένα ποιος κάνει τι και ποιος είναι ο ρόλος και οι ευθύνες του καθενός. Οι οργανισμοί δημιουργούνται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργικής συνεργασίας. δεν εμπλέκονται, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη νομική τους βάση διότι αυτό αντιβαίνει το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης. Δεν εμπλέκονται λοιπόν στην διατύπωση και την ανάπτυξη πολιτικής ατζέντα. Αυτή την πολιτική ημερήσια διάταξη την ορίζει την ορίζουν τα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, υπό την πρωτοβουλία της Κομισιόν, αν χρειαστεί. Αλλά φυσικά ο δημοκρατικός έλεγχος και για τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και για τις κυβερνήσεις. Ο δημοκρατικός έλεγχος λοιπόν ασκείται όταν ορίζονται αυτές οι πολιτικές ημερήσιες διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται μετά από τους οργανισμούς μέσα βέβαια από τις δικές τους αρμοδιότητες ο καθένας. Τρίτη υπόμνηση κυρίες και κύριοι βουλευτές. Εμείς Έχουμε έναν τομέα όπου υπάρχει μεγάλος καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Γι' αυτό λοιπόν είναι και ουσιαστικότατη μια πρωτοβουλία σαν αυτή που επιτρέπουν σε δύο δημοκρατικά όργανα να συνδιαλλαγούν και να θέσουν και τη βάση της συνεργασίας μεταξύ τους. Λοιπόν, παράδειγμα, τι θα συζητήσετε σήμερα το απόγευμα ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Το πολιτικό αριθμιστικό, το πολιτικό πλαίσιο, το εθνικό πολιτικό πλαίσιο, το γενικό αριθμιστικό πλαίσιο το ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κάθε κράτος είναι αρμόδιο για να εφαρμόζει την πολιτική αυτή. όσον αφορά δηλαδή το εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είναι υπό την αρμοδιότητα του κράτους. Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν πληρεί τα καθήκοντά το Frontex. Οι κοινέ δράσεις του Frontex συντονίζονται από το Frontex, αλλά την πρώτη αρμοδιότητα την έχει το κράτος μέλος, το οποίο έχει αποφασίσει και εκτελεί αυτά αυτά, αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις. Αν χρειαστεί βεβαίως μπορεί να αποφασιστεί κάτι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτάκτος. Αλλά ο δημοκρατικός έλεγχος ασκείται μέσα στο ίδιο το κράτος μέλος από τους δικούς του δημοκρατικούς μηχανισμούς. Τρίτα, τελευταίο να θυμίσω κύριε Πρόεδρε. Είπατε, πρέπει να δημιουργήσουμε μια θετική δυναμική. Είναι απαραίτητο. Απολύτως απαραίτητο θα έλεγα. Έστω και αν η ατζέντα για τα, θέματα, για τα εσωτερικά θέματα και θέματα δικαιοσύνης είναι πρόσφατα, εντυπωσιαζόμαστε από τον μεγάλο αριθμό των διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και εσείς θα εξετάσετε ήδη τρεις από αυτούς τους οργανισμούς, Frontex, Europol και Eurojust. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι τρεις δυναμικοί οργανισμοί σήμερα. Είναι ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, το ΣΕΠΟΛ για την αστυνομική κατάρτιση και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Άλλοι δυο οργανισμοί βραχυπρόθεσμα μακροπρόθεσμα θα συσταθούν. Το ΑΖΟΚ είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου το οποίο θα αρχίσει να δουλεύει στα τέλη της χρονιάς ή στην αρχή του 2011 και αν ο συνομοθέτης αποφασίσει το, ο μελλοντικό οργανισμός για τη διαχείριση των μεγάλων ε, πληροφοριακών συστημάτων. Δηλαδή κάπου 8 οργανισμοί πολλοί οργανισμοί. Αλλά ο τομέας της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων είναι το ε, τομείς όπου η λειτουργική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη δηλαδή των διαφόρων πολιτικών θέσεων και την εφαρμογή τους. Είναι λοιπόν απόλυτα λογικό. Φυσικά βέβαια όταν πληρούνται όλοι οι νομικοί και δημοκρατικοί όροι να προσφεύγουμε σε οργανισμούς οι οποίοι είναι οι, οι δήμονες για την υποστήριξη και την οργάνωση αυτής της λειτουργικής συνεργασίας. Η θετική δυναμική που αναφέρατε εσείς κύριε Πρόεδρε είναι εφικτή, υπάρχει. Παράδειγμα, το άλλο θέμα που θα συζητήσετε αύριο, η συνεργασία στα πλαίσια του Σέγγεν. Και να το δω λίγο πιο μακροπρόθεσμα το θέμα. Μέχρι να ισχύσει η συνθήκη του Άμστερνταμ, η συνεργασία Σέγγεν ήταν μια διακυβερνητική συνεργασία, στενά διακυβερνητική. Μερικοί είπανε ότι επρόκειτο και για, το εργαστήριο της μελλοντικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λάμβανε χώρα εντελώς έξω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από διάφορα ψηφίσματα αναφέρθηκε πολλές φορές για το Σέγγεν και ο τόνος αυτός των ψηφισμάτων ήταν σαφής. πρόκειται για μια απόρριψη και μια πολύ σκληρή κριτική. Άρχισε να ισχύει το Άμστερνταμ και η Λισαβόνα ισχύει σήμερα. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν ότι όλα τα θέματα τα οποία κατέστησαν κοινοτικά μετά το Άμστερνταμ και τα οποία αφορούν στο κεκτημένο του Σέγγεν ελέγχονται σήμερα απόλυτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο ορίστηκε μέσα από συναπόφαση. Είτε για τον κοινό κώδικα για το πέρασμα των εξωτερικών συνόρων, είτε για τον κοινό κώδικα για τη χορήγηση της θεώρησης της βίζας είτε για το κεκτημένο CS2 είτε για τη νομική βάση του TVS και για να μην αναφέρω κι άλλα όλα αυτά τα νομικά μέσα τα οποία εμείς έχουμε κληρονομήσει από το κεκτημένο του Σέγγεν και τα ανέπτυξε το κεκτημένο του Σέγγεν έχουν συναποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει λοιπόν αυτή η δυναμική θετική δυναμική. Πολλά πράγματα ήδη έχουν γίνει και πολλά πράγματα είναι και δυνατά να γίνουν στα πλαίσια δηλαδή των μέσων που έχουμε σήμερα. Εσείς είστε συνομοθέτες, θυμηθείτε το. Η μεταρρύθμιση για παράδειγμα του Frontex. Αποφασίσατε εσείς τη νομική βάση του Frontex. Αποφασίσατε τη δημιουργία των Rabbits των ομάδων ε, γρήγορης επέμβασης. Ο κύριος Μπουσουτήλ ήταν εισηγητής. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τεράστιες αρμοδιότητες ως συνομοθέτης. Επίσης είστε και δημοσιονομική αρχή. Είστε αρχή του προϋπολογισμού. Όλα λοιπόν τα όργανα αυτά χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και εσείς λοιπόν έχετε τεράστιες δυνατότητες ως όργανο προϋπολογισμού να ορίζετε τη χρηματοδότηση αυτών των οργάνων. Επίσης, η βάση, η ιδρυτική βάση αυτών των οργανισμών προβλέπει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του reporting. Η Europol, ας πούμε, άρθρο 47, αν θυμάμαι καλά ότι η Ευρωπολή έχει αυτή την υποχρέωση. Αλλά και σε άλλα κείμενα, τα συστατικά κείμενα δηλαδή τα ιδρυτικά συγγνώμη, κείμενα των διαφόρων οργανισμών διαπιστώνατε ότι αυτή υπάρχει υποχρέωση. Και εσείς ως Εθνικά Κοινοβούλια μπορείτε να καλείτε όποτε θέλετε τους γενικούς διευθυντές αυτών των οργανισμών να έρχονται να σας τα λένε. Και ελάχιστοι εκτελεστικοί διευθυντές θα αρνιόντουσαν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια πρόσκληση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο. Ο κύριος Κούκελμπερκ ανέφερε την ανακοίνωση που θα παρουσιάσει τον Νοέμβριο η Κομισιόν για τα, τις ε, λειτουργικές πλευρές της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Φυσικά θα επανέλθουμε στο θέμα και θα το δείτε κι εσείς και πάλι θα επανέλθετε. Αλλά η Κομισιόν έχει την πρόθεση να προτείνει διαδικασίες για το policy cycle. Καλά κάνετε και το λέτε αγγλικά γιατί αν το λέγαμε γαλλικά θα ήταν πολύ μακρύτερος ο όρος. Και αυτό το policy cycle θα επιτρέπει το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στον καθορισμό των προαιρεοτήτων αυτής της στρατηγικής, να την αξιολογεί κτλ. Εξού λοιπόν και η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει, να είναι παρόν όταν εκφράζονται αυτές οι πολιτικές επιλογές και όταν μετά θα εφαρμόζονται από τους οργανισμούς. Αναφέρατε κύριε Πρόεδρε και τις ανησυχίες του σώματος για το δημοκρατικό έλεγχο επί της Ευρωπόλ. Η κυρία Μένστρομ ε, είχε την ευκαιρία να εκφραστεί σχετικά πολλές φορές. Για το νομικό πλαίσιο δηλαδή της Europol έχουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη της χρονιάς. Πρόκειται για κάτι το μακροπρόθεσμο και μακρόπνοο. Ε, αυτό θα προχωρήσει και μέσα από την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της νέας απόφασης του Συμβουλίου είναι σαφώς, σαφές όμως ότι η ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου δεν μπορεί να περιμένει. Έχουμε ακόμη πολλά που θα λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της Europol. Δεν είναι μια αστυνομική υπηρεσία, δεν έχει λειτουργικές αρμοδιότητες, δεν έχει ανακριτικές δυνατότητες. Επίσης η Europol βασίζεται στην στενή συνεργασία με τις εθνικές αστυνομίες. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνει ένα συνδυασμός εθνικού δημοκρατικού ελέγχου και ευρωπαϊκού δημοκρατικού ελέγχου. Αυτά η Κομισιόν Φυσικά είναι αυτονόητο ότι εμείς είμαστε όλοι αυτοί να ακούσουμε τι θα μας πείτε σε αυτές τις επόμενες ώρες εργασίας για να βρεθεί μια καλύτερη συντονιστική λύση Πολλές φορές τα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν έγκαιρα τις πληροφορίες που τους χρειάζονται για να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους του δημοκρατικού ελέγχου. Και αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελεί και ένα κεκτημένο αυτών των σημερινών σας εργασιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ένα διήμερο σεμινάριο. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου το χρόνο για να καλύψουμε όλα μας τα θέματα. Έχουμε ε, δύο συνόδους εργασίας σήμερα το απόγευμα. Η πρώτη σχετίζεται με την Frontex, η δεύτερη με την Europol. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε κατευθείαν ε, στο πρώτο μέρος, μετά από το οποίο θα δώσουμε το λόγο ε, στους αντιπροσώπους ε, για συζήτηση και θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων που βρίσκονται στην αίθουσα καθώς και στα μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα καλέσω λοιπόν τον κύριο Ιλκα Λατίνεν που είναι ο Διευθυντής της Frontex Simon Bosutil. τον Σάιμον Μποσούτιλ που είναι η συγητής για αναθεώρηση της εντολής της Frontex, μέλος της Επιτροπής Λίμπε και συντονιστής. Και τον κύριο Άντρεϊ Μούνκο που είναι μέλος ε, του ε, Γερμανικού ε, Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που σας βλέπω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το πρώτο αυτό μέρος ε, της ε, συζήτησης ε, για την υπηρεσία Frontex. Πρώτος που θα πάρει το λόγο θα είναι ο κύριος Ιλκα Λατίνεν που είναι Διευθυντής της υπηρεσίας Frontex. Κύριε Λατίνεν, καλώς ήρθατε. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ε, συζήτηση αυτή που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα ποτέ δεν είναι στατική. Παρότι μέχρι τώρα είχαμε, φέτος είχαμε ε, μείωση της ε, παράτυπης μετανάστευσης κατά 20% σε σχέση με πέρσι, έχουμε δει και αύξηση της ε, συγκέντρωσης των οδών καθώς αυτοί που διευκολύνουν το παράνομο πέρασμα των συνόρων συνεχίζουν να ε, βρίσκουν νέους, νέες ε, οδούς. Ε, καθότι οι, οι ομάδες χρησιμοποιούσαν διαφορετικές οδούς στο παρελθόν, ενώ τώρα έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Μετά από το πρώτο εξάμεινο της φετινής χρονιάς η οδός αυτή ε, αντιπροσωπεύει το 80% των ε, παράνομων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είναι τώρα η βασική χώρα διέλευσης ε, για λαθρομετανάστες που προορίζονται για την Ευρώπη. Συνήθως πετάνε στο Ίστανπουλ λαθρομετανάστες και μετά περνάνε τα χερσαία σύνορα. Μία από τις βασικές τροποποιήσεις στο σύνορο αυτό ήταν η μεταφορά από τη θάλασσα στην, ε, στη Στεριά. Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ε, ε, Ποσειδών 2010 επικεντρωνόμασταν στα θαλάσσια σύνορα ενώ τώρα μεγαλύτερη πίεση βλέπουμε στα χερσαία σύνορα 73% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010. Αλλού η κατάσταση είναι πολύ λιγότερο δραματική από ό,τι σε προηγούμενα έτη. Κάποτε η περιβόητη οδός Δυτικής Αφρικής από την ε, Σενεγάλη και τη Μαυριτανία στα Κανάρια νησιά τώρα έχει ε, κλείσει σχεδόν τελείως ε, λόγω του, της επιχείρησης Ήρα, της πρώτης επιχείρησης Frontex και η οποία συνεχίζεται ακόμα. Οι κοινέ επιχειρήσεις Μινέρβα, Ιντάλλο και Ερμής συνεχίζουν να μειώνουν την λαθρομετανάστευση στην ε, Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο. Και το πρόγραμμα Ποσειδών, όπως είπα, έχει κλείσει μεγάλο μέρος ε, των μετακινήσεων στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Ε, Η βασική πρόκληση τώρα βρίσκεται στα χερσαία σύνορα. Όσον αφορά τα άλλα χερσαία σύνορα, ε, τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας ε, και της Λευκορωσίας ε, παραμένουν γενικά σταθερά, ενώ η κατάσταση στα σύνορα Ουγγαρίας-Σερβίας ε, αποτελεί ε, συνέχεια της κατάστασης, ε, στην Νότια Ελλάδα. Οι λαθρομετανάστες κινούνται βόρεια προς τις χώρες προορισμού τους, περνάνε από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Σερβία με στόχο να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα σύνορα της Ουγγαρίας. Αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει με την μελλοντική προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο Σέγγεν η αλλαγή των εξωτερικών συνόρων ε, δεν θα ε, διπλασιάσει μόνο το μήκος των ε, χερσαίων συνόρων με την Τουρκία απαλλάσσοντας έτσι την Ελλάδα από μέρος της πίεσης αλλά θα δημιουργήσει και ένα σαφές πέρασμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα έχει περάσει κάποιος τα εξωτερικά σύνορα. Έχουμε δει αυξημένη δραστηριότητα στα βουλγαρικά σύνορα, αλλά είναι πολύ νωρί να πούμε αν αυτό αποτελεί μόνιμη τάση. Κύριε Πρόεδρε, όπω είπα στην αρχή, η κατάσταση στα σύνορα ποτέ δεν είναι στατική. Χρειάζεται ε, επικαιροποιημένε πληροφορίε, ε, μια ολοκληρωμένη στρατηγική και μια ευέλικτη προσέγγιση. Ε, όλα αυτά στα πλαίσια τη ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων IBM. Το, η σημασία ε, του IBM ε, ε, ε, εμπλουτίστηκε πριν ε, πρόσφατα με την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει αχρηστική γραμμή ανάμεσα στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα. Το IBM έχει γίνει ένα απαραίτητο κομμάτι της εσωτερικής στρατηγικής ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Το στοιχείο που λείπει είναι να διαγράψουμε τα διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους πυλώνες στο μυαλό μας μέσα. Η ασφάλεια των συνόρων ε, ε, ε, είναι κάτι που απαιτεί πάνω από μία υπηρεσία και δεν υπάρχει μία υπηρεσία που να μπορεί ε, να ελέγξει το, τη ροή των επιβατών στα σύνορα οι συνοριακές ε, αρχές, ε, τα τελωνία, η αστυνομία, οι αρχές μετανάστευσης και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους. Έχοντας λοιπόν κατά νου την νέα νομική κατάσταση, ε, έλεγχοι των συνόρων θα πρέπει να μπορούν να γίνουν οπουδήποτε υπάρχει έλεγχος της ροής των επιβατών. Αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιο προξενείο σε τρίτη χώρα, όπου εκδίδονται βίζες ή σε κάποιο αεροδρόμιο στο έδαφος της Ευρωπαϊ... κάποιο κράτους μέλος. Επίσης, ε, Υπάρχουν πολλέ περιπτώσεις όπου οι αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ε, θέλουμε ε, οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση. Αυτό είναι κάτι που ε, αγωνίζεται η υπηρεσία μας να το πετύχει κάθε μέρα. Στόχος, ο τελικός μας στόχος είναι να μειωθεί η ροή των λαθρομεταναστών για να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι συνθήκες Λισαβόνα και το πρόγραμμα Στοκχόλμης έχουν επιφέρει επίσης μια άλλη σημαντική αλλαγή. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχουν ε, μπει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η πρόκληση εδώ είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν την πρόκληση ε, να κάνουμε τα σύνορα της Ευρώπης ε, περατά από τους ε, από την μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιωτών, των νόμων ταξιδιωτών, παρέχοντας όμως και την ασφάλεια που τους αξίζει. η καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρώπων και της λαθρομετανάστευσης ε, απαιτεί και ανθρώπους και δυναμικό. Όσον αφορά τις ε, λεπτομέρειες αυτών που θα ήθελα να δω στον αναθεωρημένο κανονισμό Frontex, μπορώ να είμαι συγκεκριμένος. Πρώτον, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για να καταπολεμήσουμε τις ε, απειλές προς τις αξίες μας όπως είναι η εμπορία των ανθρώπων, ιδιαίτερα η πώληση και μεταφορά ανθρώπων, συχνά ανηλίκων ε, για ε, σεξουαλική κακομεταχείριση ή την, πώληση οργάνων για, για θα πρέπει να μπορούμε να ελέγχουμε τα ονόματά τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ό,τι στοιχεία έχουμε για να έχουμε καλύτερα στοχευμένες επιχειρήσεις στα σύνορα. 400.000 συνοριοφύλακες ε, θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην ε, καταπολέμηση του ε, εγκλήματος και των εγκληματικών οργανώσεων στα σύνορα. Μας ε, ενδιαφέρει να εντοπίσουμε τους ε, ανθρώπους που κινδυνεύουν ε, από τα εγκλήματα των εγκληματικών οργανώσεων. Όταν υπάρχουν στοιχεία, όταν υπάρχουν υποψίες για οργανωμένο έγκλημα και ε, όποιος έχει τα στοιχεία αυτά δεν ε, τα υποβάλλει στην ε, Europol δείχνει πόσο ανεπαρκές είναι το σύστημα. Οι πληροφορίες αυτές συχνά παραμένουν σε τοπικό επίπεδο όπου δεν χρησιμεύουν. Μια τέτοια κατάσταση εξυπηρετεί ε, τα συμφέροντα του οργανωμένου εγκλήματος ε, εις βάρος της ε, πρόληψης του εγκλήματος και της προστασίας των θυμάτων. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ολιστική διπηρεσιακή προσέγγιση στην καταπολέμηση του εγκλήματος εάν οι πολύτιμες πληροφορίες παραμένουν σε τοπικό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, Επίσης μας απασχολεί η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, τα κράτη-μέλη διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό ε, στην Frontex σε θελοντική βάση, ε, αλλά για να υπάρχει αποτελεσματικός προγραμματισμός και επιχειρησιακή διαχείριση θα πρέπει να έχουμε εγγυήσει ότι θα παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι στους ε, σωστούς ανθρώπους ε, τη σωστή στιγμή. Επικροτούμε την πρόταση της Κομισιόν να δημιουργήσουμε ε, μια, μια πηγή τεχνικού εξοπλισμού με ισχυρότερη δέσμευση από τα κράτη-μέλη και θα θέλαμε περισσότερη βεβαιότητα έχοντας εξοπλισμό που να είναι η ιδιοκτησία της Frontex ή η συνειδιοκτησία. Αυτή η αυξημένη ευελιξία και αυτονομία θα βελτιώσει τη δυνατότητά μας να ε, διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους ε, πόρους και θα μειώσει τον χρόνο αντίδρασής μας ε, και θα βελτιώσει την προσαρμογή μας στην κατάσταση που αλλάζει συνεχώς. Αλλά πιο σημαντικό μα πόρο δεν είναι τεχνικό. Οι καλύτερε πληροφορίε, ο καλύτερο προγραμματισμό και οι απαραίτητοι πόροι ε, δεν αξίζουν τίποτα αν δεν υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι. Και αυτή αποτελεί μια από τι σημαντικότερε συμβολέ ε, των κρατών μελών. Οι συνοριοφύλακε και άλλοι εμπειρογνώμονε. Ε, και θα ήθελα εδώ να πω ότι θα ήθελα αυξημένο δυναμικό οι αποσπασμένοι ε, εθνικοί ε, αξιωματικοί θα ενισχύσουν την ε, μας, το επιχειρησιακό μας δυναμικό και θα διασφαλίσουν συνέπεια και συνέχεια όχι μόνο στις επιχειρήσεις της Frontex αλλά και στην συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πάλι οι λέξεις κλειδιά είναι αυτονομία και ευελιξία. Και τέλος, αλεξίσου σημαντικό, Υπάρχει το θέμα της ε, συνηγεσίας. Για να βελτιώσουμε το επιχειρησιακό προφίλ της Frontex, ε, να μην είναι απλά συντονιστής, αλλά να είναι ε, συνηγέτης μαζί με το κράτος μέλος υποδοχής μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, θα πρέπει... αυτό θα ήταν προς όφελος του συνόλου της Ευρώπης. Η αυξημένη αλληλεγγύη και η αίσθηση μοιρασμένης ευθύνης είναι απαραίτητη ε, για την αποστολή της Frontex να δημιουργήσει την αίσθηση μοιρασμένη ευθύνη, αμοιβαίας ε, εμπιστοσύνη ε, που θα, στηρίζει, που θα δείχνει την πραγματική αξία των κοινών επιχειρήσεων. Κύριε Πρόεδρε, το δικαίωμα να ε, διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα ανθρώπων που αποτελούν ε, πιθανή απειλή στην ασφάλεια της Ευρώπης και, και, τους, και τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας, αυτό είναι απαραίτητο. Η δυνατότητα συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι απαραίτητη για να πετύχουμε τους στόχους του προγράμματος της Στοκχόλμης. Θέλουμε συνειδιοκτησία, συνδιαχείριση, ε, συνηγεσία και συνεργασία. Το ε, μήνυμα είναι σαφές, θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γάτινεν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προτείνω να, προτείνω να προχωρήσουμε με τον εισηγητή της εντολής Frontex, Simon Μπουσούτη, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά προτείνω επίσης για να επαρκέσει ο χρόνος και για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα εργασίας μας ε, έγκαιρα, χωρίς καθυστερήσεις, να μπορέσουμε να περιοριστούμε σε 10 λεπτά ώστε να ξεκινήσει μετά η συζήτηση. Κύριε Μπουσούτιλ, έχετε τον λόγο λοιπόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, μεγάλη χαρά είναι για μένα να είμαι εδώ και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που μπορώ να έχω αυτή την ευκαιρία να έχω μια ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους μας, ιδιαίτερα από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η συγκυρία και η χρονική αυτή συγκυρία δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη για αυτή την κοινοβουλευτική συνεδρίαση. Είχαμε πρόσφατα μία πενταμελή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήγε στη Βαρσοβία και να επισκεφθεί τον κύριο Λάιτενεν και την ομάδα του Frontex. Και έχουμε σήμερα αυτή την ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων. Ω εισηγητή για αυτό το χαρτοφυλάκιο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πρόθεσή μα να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το χαρτοφυλάκιο ήδη την επόμενη εβδομάδα. Η χρονική συγκυρία λοιπόν αυτών των συνεδριάσεων μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη στη σύμπτωση αυτή. Θα περιοριστώ να διατυπώσω έξι ερωτήματα ή θέματα που ελπίζω εγώ ως εισηγητής ότι θα μπορέσετε εσείς να με βοηθήσετε να τα απαντήσω έγκαιρα ώστε να προετοιμάσω έγκαιρα την έκθεσή μου και τις τροπολογίες για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Θα προσπαθήσω μόνο σε ένα από αυτά τα ερωτήματα να απαντήσω λόγω περιορισμένου χρόνου φυσικά και θα σας αφήσω εσάς την μεγάλη πλήρη χαρά να απαντήσετε τα υπόλοιπα πέντε ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να διατυπώσω και θα ήθελα εμείς να ερωτηθούμε γι' αυτό είναι πού στοχεύει και πού κατευθύνεται η Frontex σήμερα. Γενικό αυτό, λόγο έτσι δεν είναι, αλλά πρέπει να έχουμε μια πολιτική συζήτηση για το τι θα θέλαμε εμείς για να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, τι θα θέλαμε να είναι η Frontex όταν ενηλικιωθεί, όταν μεγαλώσει. Πέντε χρόνια λειτουργεί, έξι χρόνια μετά τον κανονισμό της. Έχει μία πείρα πέντε ετών. Πού θέλουμε λοιπόν αυτό ο οργανισμός να πορευθεί να οδεύσει προς το μέλλον. Αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατυπώσουμε και να απαντηθεί. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια χαλαρή συνεργασία μεταξύ μας όταν έρχεται η στιγμή να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα ή θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη, πλήρως ολοκληρωμένη και μια πλήρως ευρωπαϊκή υπηρεσία φύλαξης σύνορων. Δεύτερο ερώτημα σε ποιους τομείς και παιδεία θέλουμε η Frontex να δραστηριοποιείται και να είναι πιο αποτελεσματική. Σαφές είναι ότι τα πρώτα έτη εμπειρίας έδειξαν ότι η Frontex ήταν επικοδομητική και θετική στη λειτουργία της σε κάποιους τομείς, λιγότερο αποτελεσματική σε άλλους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτή τη νέα νομοθετική διαδικασία τη Frontex να είναι πιο αποτελεσματική. Πρέπει εκεί να δώσουμε input, να δώσουμε προτάσεις σε κοινέ δράσεις, joint operations και πώς σε επιστροφές ατόμων, σε ε, επανεισδοχή ε, όσον αφορά τρίτες χώρες, ίσως είναι τομείς που θα έπρεπε να τις εξετάσουμε από πιο κοντά για να είναι πιο αποτελεσματική υπηρεσία. Το τρίτο ερώτημα που θα ήθελα να διαρωτηθούμε και να μας απασχολήσει συσχετίζεται με την συσσόρευση και στελέχωση συνοριοφυλάκων. Ξέρουμε ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα η Frontex για να βοηθήσει τους συνοριοφύλακες να συνέρχονται και κυριολεκτικά να κατανοούν ο ένας τον άλλο και ακόμα και να ακολουθούν μια κοινή οδό κατάρτισης ε, και εκπαίδευσης. Αυτό είναι καινούριο και έγινε χάρη στη Frontex τα τελευταία χρόνια. Τώρα όμως βλέπουμε και παρακολουθούμε και διαπιστώνουμε ότι έχει μια ομάδα έκτακτης δράσης, rabbits, για επίγουσες δράσεις, της rabbits. Δεν είναι ο καλύτερος όρος, αλλά υπάρχει λοιπόν αυτή η μονάδα rabbits. Και έχουμε επίσης και ειδικέ ομάδες υποστήριξης και συνδρομής για κοινέ δράσεις, τις κοινέ ομάδες της Frontex. Πού θέλουμε να πορευθούν όλες αυτές. Θέλουμε να προχωρήσουν και σε ποιο εύρος και βαθμό θέλουμε να συσσωρευθούν, να γίνει ένα πουλ και να υπάρξουν συνοριοφύλακες διαφορετικών κρατών μελών σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο που θα δρουν. Τέταρτη ερώτηση που θα ήθελα να μας απασχολήσει και αυτή συσχετίζεται πάλι σε pooled resources, σε συσσωρευμένους από, κοινού <clears throat> ε, συνοριοφύλακες και υλικό και εξοπλισμό. Πώς θα διασφαλίσουμε όλα τα κράτη-μέλη να συνδράμουν και να κάνουν αυτό το οποίο είναι αναγκαίο ώστε να υποστηρίξουν την Frontex από πλευρά στελεχών και υλικού και εξοπλισμού. Ξέρουμε ότι δεν έκαναν αρκετά μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να τα πείσουμε και να τα κινητοποιήσουμε να συμμετάσχουν περισσότερο και πώς μπορούμε ουσιαστικά να οδηγήσουμε στο να λειτουργεί αλληλεγγύη στην πρακτική καθημερινή μορφή και δράση. Και το επόμενο ερώτημα και συσχετίζεται με τα, όσα είπε ο κύριος ε, Λάιτινεν. Προσωπικά δεδομένα. Θα έπρεπε η Frontex να είναι σε θέση να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων για να μπορεί να καλύψει τις δράσεις και το έργο της πιο αποτελεσματικά και να είναι πιο αποτελεσματική, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση του εγκλήματος, διασυνοριακού, διεθνούς εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης. Και τέλος, εν τέλει, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε η ε, Frontex να λογοδοτεί περισσότερο σε εμάς στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Α χρησιμοποιήσω τα υπόλοιπα 4,5 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου για να καλύψω αυτό το τελευταίο ερώτημα της δημοκρατικής λογοδοσίας. Θα ήθελα να χωρίσω αυτό το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος, λογοδοσία κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Και τυχαίνει να είμαστε σε αυτή τη στιγμή στο νομοθετικό έργο, διότι καθώς γνωρίζετε τροποποιούμε τον κανονισμό αυτή τη στιγμή λειτουργίας ε, της Frontex. Είναι σαφής ο ρόλος για σας συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είχατε την ευκαιρία να ε, εκφράσετε τις απόψεις σας. Μετά από την προθεσμία των 8 εβδομάδων, έξι <clears throat> σώματα από τα Εθνικά Κοινοβούλια υιοθέτησαν γνωμοδότηση και είχαμε τεκμηριωμένη γνωμοδότηση από τη Γερουσία της Πολωνίας που μας είπε ότι δεν είναι συμβατή αυτή η πρόταση με την αρχή της, της επικουρικότητας. Η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή φυσικά που μέσα σε αυτήν συνερχόμαστε σήμερα είναι μια άλλη καλή ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι θα αυξηθεί η λογοδοσία, δημοκρατική λογοδοσία αυτής της υπηρεσίας είναι εξαιρετική ευκαιρία που έχουμε να έχουμε τον εκτελεστικό διευθυντή εδώ της υπηρεσίας και να μπορέσουν να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα με αυτόν τον τρόπο. Στην στο νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου πάλι έχουμε ένα συγκεκριμένο χειροπιαστό τομέα, ένα πεδίο όπου μπορεί να ασκηθεί η δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά την υπηρεσία. Διότι εμείς θα προτείνουμε τις τροπολογίες μας με βάση το feedback και τις απαντήσεις και τοποθετήσεις που θα έχουν ε, υπάρξει από την υπηρεσία. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ένα επεισόδιο το οποίο συνέβη νωρίτερα εφέτος στην Ευρωβουλή όταν είχαμε την ούτως αποκαλούμενη ε, τις ούτως αποκαλούμενες κατευθυντήριες γραμμές Frontex, Frontex Guidelines, που είχαν προταθεί σε σχέση με την επιτροπολογία στο Ευρωκοινοβούλιο. Πράγμα το οποίο σήμαινε ότι εμείς ως ε, θεσμικό όργανο θα μπορούσαμε ή να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το σύνολο των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών, Guidelines, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε το ένα ή άλλο. Αυτό το ε, στοιχείο, αυτό το θέμα κατέληξε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο 10. Προσέφυγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Διότι θεώρησε ότι δεν ήταν αυτή η σωστή διαδικασία. Η σωστή διαδικασία θα έπρεπε να είναι η διαδικασία συνομοθέτη. Συνομοθετικό έργο που θα είχε δυνατότητα να αυξήσει τι αρμοδιότητε του Ευρωκοινοβουλίου. Πρώτο σκέλο αυτό. Δεύτερο σκέλο. Να δούμε πώ μπορούμε να αυξήσουμε την δημοκρατική λογοδοσία μετά την ε, ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό. Παράδειγμα, κάθε χρόνο το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας να ζητήσουμε από τις υπηρεσίες και οργανισμούς, την Frontex και άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες, τι ακριβώς κάνουν και πώς το κάνουν. Προτού δώσουμε νέα κονδύλια ή εγκρίνουμε νέα κονδύλια ή κιόλας αυξήσουμε και τα κονδύλια τους στον προϋπολογισμό. Δεύτερον, κάθε χρόνο χορηγούμε απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπου λέμε ότι χρησιμοποιήθηκε αποτελεσματικά ο προϋπολογισμός με τα κονδύλια του από τις υπηρεσίες ή όχι. Και έχουμε έχουμε και συνάδελφο που μπορεί να μας πει πολλά για αυτό το θέμα. Και είναι ένα μέσο, ένας μοχλός στα χέρια μας που μπορούμε με αυτό να αυξήσουμε την δημοκρατική λογοδοσία των υπηρεσιών και ε, οργανισμών. Θα πρέπει να μας υποβάλουν έκθεση, να προσέρχονται εδώ και να παρουσιάζουν αυτά τα στοιχεία και κάθε υπηρεσία και οργανισμός παρουσιάζει και ένα πρόγραμμα εργασίας προηγούμενα, πριν δηλαδή εγκριθεί ο προπολογισμό για το επόμενο έτος. Και αυτή είναι πάλι άλλη μια ευκαιρία να διατυπώνονται ερωτήματα. Και εδώ πάλι έχουμε την ευκαιρία και για άλλους οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, τον επόπτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι απόψεις αυτού και των άλλων μπορούν να μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την ε, δημοκρατική λογοδοσία. Έχω μόνο 10 δευτερόλεπτα βλέπω στη διάθεσή μου. Θα ολοκληρώσω λοιπόν. Δεν ολοκληρώσα, δεν συμπεριέλαβα όλα όσα ήθελα να πω, αλλά θα συμπεριλάβω αυτό το σημείο. Αν κάποιο από εσά έχει κάποια πρόταση ως feedback που θέλει να μου διαθέσει, να μου δώσει, παρακαλώ μέσω της ιστοσελίδας ε, του Κοινοβουλίου να μου το αποστείλει. Θα ολοκληρώσω την έκθεσή μου και με μεγάλη χαρά θα λάβω προτάσεις σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ για την παρέμβασή σας και σας ευχαριστώ που τηρήσατε με τέτοια ακρίβεια τα 10 λεπτά που σας είχαν δοθεί. Τώρα περνάμε στον κύριο Χόγκο, εκπρόσωπο του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να μιλήσω σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες επικρίσεις για τη Frontex. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Επιχειρησιακή Συνεργασία στα Εξωτερικά Σύνορα, Frontex, από την ίδρυσή της το 2004, έχει ε, ε, αποτελέσει επίκεντρο πολλών επικρίσεων. Και ο λόγος ε, για την κριτική αυτή είναι η ανθρώπινη τραγωδία που εκτιλήσεται στα εξωτερικά σύνορα. Ξέρετε τα νούμερα, 10.000 άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν ε, πεθάνει. Ε, και εδώ στην, ε, στις Βρυξέλλες πέρσι έγινε διαδήλωση κατά της Frontex. Θα σας αναφέρω κάποιες από αυτές τις επικρίσεις. Πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τα μέτρα της Frontex στην Μεσόγειο. Ιδιαίτερα το ότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία των ε, προσφύγων. Μια γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συνοριοφύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενεργούν και εκτός των συνόρων, ε, δηλαδή ε, πέρα από το όριο των 12 μιλίων. Οι πρόσφυγες που, που πιάνονται στη θάλασσα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουν πέρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την μεταχείριση των προσφύγων σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει εμεί ω ε, βουλευτέ να φροντίσουμε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα αυτά δικαιώματα και η προστασία των ε, προσφύγων. Και έτσι φτάνω στο επόμενο, ε, στην επόμενη επίκριση. Με βάση αυτή την ανεπαρκή προστασία των προσφύγων, τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τα σχέδια τη ευρωπαϊκή Ένωση για τη Frontex όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, είναι μάλλον ύποπτα. Εδώ τίθεται το θέμα τη επικουρικότητα. Υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια που συμφωνούν. Και σκέφτομαι για παράδειγμα την έκθεση του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει ε, να σταματήσουμε την, ε, τις εξελίξεις αυτές. Το να γίνει η ε, Frontex μια σούπερ υπηρεσία για την, απομάκρυνση των προσφύγων, αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Αυτό θα ήταν παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα οδηγήσει σε αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την τακτική σαλάμι, το να κόβουμε τα πράγματα σε μικρά κομμάτια, δίνουμε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες ε, στην υπηρεσία αυτή παρακάμπτοντα τι συνθήκες. Και έτσι φτάνω στην τετρίτη βασική επίκριση, ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς επαρκή δημοκρατικό έλεγχο και αυτό έχει αναφερθεί. Ακριβώς επειδή στα πλαίσια της Frontex ε, η διακυβερνητική συνεργασία έχει, σημαντική, έχει μεγάλη σημασία. Τίθεται το θέμα του ελέγχου όχι μόνο με, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως η Frontex όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας για την Europol και την ε, Eurojust ε, η Frontex να λογοδοτεί απευθεία και στα εθνικά κοινοβούλια. Το ερώτημα είναι σε ποιο διοργανικό πλαίσιο θα μπορούσε να ενσωματωθεί ο έλεγχος αυτός ή μήπως Ε, μήπως να χρησιμοποιήσουμε τους εθνικούς φορείς για έλεγχο της Europol. Χρειαζόμαστε ενίσχυση των, ε, του, της δυνατότητας ελέγχου των εθνικών φορέων. Δεδομένων των ε, καθημερινών αποτυχιών της ε, Frontex στην προστασία των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν το ε, κρύβω αυτό, θα ήθελα ήδη σήμερα να καταργηθεί η Frontex, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μια μεγάλη υπηρεσία που να μην υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και θέλουμε να αναρωτιόμαστε εάν αυτές οι τακτικές τη Frontex συμφωνούν με, μια, με τις αρχές μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι αφοσιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μήπως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε μια αναθεώρηση της ε, πολιτικής απομόνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική απομόνωση αυτή δεν είχε ήδη αρκετά θύματα και Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχουμε θεμελιώδη τροποποίηση της πολιτικής προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται φορείς όπως η Frontex να συμβάλλουν ε, ώστε να ε, καταργεί το δικαίωμα των ανθρώπων να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τα αιτήματα αυτά των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε την τήρηση, το σεβασμό των ανθρώπων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, αλλά να δημιουργούμε εμεί ένα καθεστώ το οποίο να μην τηρεί ούτε τα ελάχιστα πρότυπα. Ακόμα και αν η Frontex είναι μόνο μία υπηρεσία εφαρμογή σε μια λάθο πολιτική, δεν υπάρχει λόγο να ενισχύσουμε αυτήν τη λάθος πολιτική. Να σας θυμίσω ότι οι, ε, οι πόροι που δίνονται στην Frontex τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί από 19 εκατομμύρια σε 88 θα πρέπει λοιπόν ε, η Frontex να υπόκειται σε καλύτερο ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο και γι' αυτό περιμένω σημαντικά αποτελέσματα από τη κοινοβουλευτική αυτή συνάντηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, έχω χαρίσει ένα δίλεπτο παραπάνω στην συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χούγκο. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις ακούσαμε, όχι μόνο στη φύση τους ε, και στο περιεχόμενο, αλλά και διαφορές ως προς την πολιτική προοπτική. Ο κύριος Λαϊτίνεν εκπροσωπεί ε, ένα ευρωπαϊκό όργανο, το, ο κύριος Ποσούτιλ εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και, έχουμε και εκπρόσωπο από ένα εθνικό κοινοβούλιο, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Θα δώσουμε τώρα το λόγο σε εσά. Κάποιοι βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Προτείνω όμως όλοι να περιορίσετε το χρόνο σας ώστε να έχουμε μια όσο γίνεται ευρεία συζήτηση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Άνδριου Καλαζεύσκη, ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Κυρία. Κυρία ή κύριος. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Μπουσούτιλ ρώτησε, έθεσε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πού κατευθύνεται ή πού θα πρέπει να κατευθύνεται η Frontex. Θα ήθελα να απαντήσω σύντομα, εν συντομία αυτό το ερώτημα. Φυσικά η προστασία των συνόρων μας συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι υπό την αποκλειστική αιγίδα των κρατών μελών ως εγχείρημα. Πιστεύω ότι η Frontex θα πρέπει να είναι μια επικουρική, ένας επικουρικός οργανισμός σε αυτή τη σύνδρομη. Οι δράσεις της Frontex δεν θα πρέπει να μεταφράζονται σε κάποια κράτη-μέλη ώστε να αισθάνονται ότι α, εξαιρούνται αυτά από την συμμετοχή στην προστασία των ε, εξωτερικών συνόρων μας. Έτσι βλέπω εγώ το μέλλον της Frontex ότι έτσι θα έπρεπε να διαμορφωθεί. Βέβαια, η διαχωριστική αυτή γραμμή είναι πάρα πολύ λεπτή όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε κράτους μέλους και φυσικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Frontex και των δράσεών της. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε σε βάθος, να εμβαθύνουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως, και στρέφαμε προς τον κύριο Μπούσουτη, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω Πιστεύω λέγω ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε με κάθε σαφήνεια επακριβώς ποια είναι η κατάσταση ακριβώς στα εξωτερικά μας σύνορα ποια είναι η κατάσταση αυτή και πώς θα αλλάξει στο μέλλον και πώς θα μεταβληθεί και αν ή όχι έχουμε επαρκείς πόρους και κονδύλια στη διάθεσή μας και στελεχειακό δυναμικό και εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις με ή χωρίς την Frontex με την Frontex ως υπεροργανισμό ή με την Frontex ως ένα ε, βοηθητικό οργανισμό ως μια ε, δυνατότητα συνδρομής ταυτόχρονα όμως ε, από την άλλη πλευρά ο κύριος Διευθυντής ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε και είπε ότι δεν γνωρίζει κανένα εκτελεστικό διευθυντή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οργανισμού που θα ειρνεί το μια πρόσκληση να προσέλθει εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και ότι όλοι θα δεχόντουσαν και θα έλεγαν ότι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω λοιπόν κύριε Διευθυντά εσείς ε, να, προσε... να προσεγγίσετε το Κοινοβούλιο και το ε, πολωνικό ας το πω έτσι ε, όργανο είναι δίπλα στην Frontex. Ίσως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα τον άλλο. Μπορούμε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε για να συνεννοηθούμε και τα, στα δύο, και τα δύο σώματα του, ε, της ε, Πολωνικής, ε, τα, τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα στην Πολωνία έχουν εκφράσει μέγιστο ενδιαφέρον όσον αφορά την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της Frontex. Yes. Floor goes to Mr. Gabriele. Ο κύριος Γκαμπριέλ Μποσκέτη, μέλος της Ιταλικής Βουλής. Un saluto a lei ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό σε εσά και σε όλους τους ομιλητές. Πιστεύω ότι είναι διπρόσωπο το Frontex. Έχει ένα πρόσωπο αυτό το οποίο ανέφερε ο, ο Πολωνός γερουσιαστής, δηλαδή το πρόσωπο της ελευθερίας του κράτους μέλους ε, για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. Και το άλλο πρόσωπο είναι ο συντονισμός ως προς τη γραμμή που πρέπει να δοθεί στα κράτη-μέλη. Μιλάμε για την οργάνωσης, ενός οργανισμού για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Το Frontex ήταν πολύ χρήσιμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μετανάστευσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι και για τα θέματα μετανάστευσης θα πρέπει να παραμείνει το Frontex αρμόδιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ενδείξεις και μέσα για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ε, για μια σωστή ένταξη, κοινωνική ένταξη των ε, μεταναστών. Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι αφήξεις ή οι αποβιβάσεις λαθρομεταναστών. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα. Στην ουσία η πρόσφατη Ιταλική εμπειρία οδήγησε στην σύναψη συμφωνίας με τη Λιβύη. Της δώσαμε και δυνατότητες της ε, Λιβύης, τους δώσαμε και πλοία για την περιπολία των παραλίων. Και αυτό μείωσε κατά 80% την αποβίβαση των παρανόμων μεταναστών στη χώρα μας. Βέβαια, δημιουργήθηκαν διάφορες προβληματικές στις οποίες αναφέρθηκε ο συνάδελφος της Λίνκε. Δηλαδή αφαιρείται η δυνατότητα από αυτούς που θα ήθελαν να ζητήσουν άσυλο να, ζητήσουν, να το ζητήσουν διότι δεν μπορούν να ζητήσουν το πολιτικό άσυλο στα ανοιχτά ούτε μπορούν να το ζητήσουν από τις λιβικές αρχές. Σίγουρα πρέπει να κατανοήσουμε και τις ε, διάφορες ε, παράλληλες ε, προβληματικές. 51 φυλακισμένοι αυτοκτόνησαν στην Ιταλία πέρυσι και το 51% των φυλακισμένων στις Ιταλικές φυλακές είναι μετανάστες. Ζητήσαμε διερμηνία στα δικαστήρια. Όχι μόνο όμως στα δικαστήρια αλλά και κατά τη φάση της εκτέλεσης της ποινής και διερμηνία επίσης και στα κέντρα διαπίστωσης. Αυτά τα προβλήματα φαίνονται άσχετα ίσως, αλλά άμα δεν λυθούν, δεν εγγιώνται την ανθρωπιστική αντιμετώπιση, ούτε και δίνουν σοβαρότητα στις πρακτικές μας οι στους επαναπατρισμούς. Και φυσικά, άμα δεν υπάρχει συνεργασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για να υλοποιήσουμε όλα όσα θέλουμε να υλοποιήσουμε σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να λάβετε υπόψη βέβαια και την κατάσταση της Ιταλίας που έχει όλα αυτά τα άπειρα παράλια τα οποία επιτρέπουν εύκολες αποβιβάσεις. Και φυσικά όλοι αυτοί οι μετανάστες δεν μένουν στην Ιταλία, πάνε παντού. Έχουν ζητήσει πάνω από 10 μέλη το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν, από εδώ και μπρο, προσπαθείτε να περιοριστείτε στα δύο λεπτά, ώστε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως για να προχωρήσουμε στο δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου αυτού. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Σας παρακαλώ κύριε Ένζιο να προσπαθήσετε να περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Θα το, θα εκτιμήσουμε όλοι. Ο κύριος Ένζιο από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Mulțumesc, domnule președinte, eh, stimați invitați, dragi colegi. Eh, în primul rând vreau să... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους έχουμε διακοινοβουλευτική συνάντηση για το θέμα αυτό. Τον καλύτερο ορισμό δηλαδή της περιοχής ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πόσο μάλλον που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αρμοδιότητες στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροποποίηση του κανονισμού Frontex. Είδα ότι διαφέρουν οι απόψεις εδώ Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στην Frontex και στα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα είναι απαραίτητη μια τέτοια συνεργασία κατά τη διάρκεια εκπόνησης των κοινών επιχειρήσεων ε, στα εξωτερικά σύνορα. Παρά το γεγονός ότι σε κεντρικό επίπεδο η Frontex λειτουργεί πολύ καλά. Σε επίπεδο κρατών μελών, στο επίπεδο κρατών μελών υπάρχει καλύτερη γνώση της κατάστασης των συνόρων. Βλέπω ότι συνεχίζεται η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να συζητάμε το θέμα αυτό, τη διασφάλιση δηλαδή των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των δράσεων της Frontex για να αποτρέψουμε και να καταπολεμήσουμε την ε, λαθρομετανάστευση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τις ε, κατηγορίες αυτές που έχουν ε, ακουστεί κατά της Frontex. Πιστεύετε ότι αιτιολογούνται ή όχι. Και καθότι είμαι εκπρόσωπος της Ρουμανίας, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Ρουμανίας στην διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων, διότι ε, έχουμε το 1 τρίτο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι πρόσφατα επισκεφτήκατε τη χώρα μας και διαπιστώσατε την ε, πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων. Από τις πληροφορίες που έχω υποθέτω ότι τα αποτελέσματα που είδατε είναι ικανοποιητικά. Πιστεύετε ότι μπορεί η Ρουμανία να αναλάβει την ε, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι πληρούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Ο κύριος Καρίδης έχει το λόγο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δύο λεπτά. Ο κύριος Καρίδης. Καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Τζαβάρα ε, τη σημερινή ε, συνάντησή μας εδώ. Είμαστε μια χώρα που αυτή την περίοδο αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ε, βιώνει με πολύ δραματικό τρόπο την παράνομη μετανάστευση. Τα στοιχεία δόθηκαν σε ένα βαθμό προηγούμενα. Στα χερσαία σύνορά μας με τα λινοργικά σύνορα τον τελευταίο χρόνο έχουμε πάνω από 700% αύξηση στους παράνομους μετανάστες. Το ίδιο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στα θαλάσσια σύνορά μας. Ε, για μας αποτελεί πολυτέλεια να συζητούμε εδώ εάν πρέπει η Ευρώπη συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει έναν αποτελεσματικό οργανισμό που θα προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα. Εμείς αυτό το θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι στην τελευταία έκθεση που υπήρξε από τις υπηρεσίες αξιολόγησης διαπιστώθηκαν πολλές αδυναμίες στο συντονισμό μεταξύ των εθνικών χωρών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στις αναλύσεις των κινδύνων, στους χώρους κράτησης. Εμείς θέλουμε ενίσχυση ως χώρα, γιατί και σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης στην οποία ζούμε, ε, όλο αυτό το κύμα των παράνομων μεταναστών δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Ε, έχει επίσης ιδιαίτερη αξία να δούμε και ορισμένα άλλα θέματα που όσο και αποτελεσματική να είναι η Frontex, αν δεν επιληθούν δεν πρόκειται να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα στην παράνομη μετανάστευση που βέβαια οι λόγοι που υπάρχει δεν είναι ώρα να τους αναλύσουμε εδώ μπορεί να είναι λόγοι πολέμου ή να είναι ε, λόγοι εσωτερικό, ε, φτώχειας που εμείς όλα αυτά τα κατανοούμε αλλά όμως ως χώρα θέλουμε να υπάρξει αποτελεσματική δράση. Ένα θέμα που υπάρχει για μας είναι το θέμα με την Τουρκία. Η Τουρκία ποτέ μέχρι τώρα δεν διασφάλισε τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και στα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και στα χερσαία σύνορα. Και εδώ πρέπει μια κουβέντα κύριε Πρόεδρε. Και εδώ πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο θέμα είναι η αλλαγή του Δουβλίνου 2. Η επανεισδοχή σε εμάς των παράνων μεταναστών αποτελεί ένα μεγάλο θέμα. Και βέβαια η στήριξη σε χώρους υποδοχής που ερχόμενοι παράνομοι μετανάστευση στην Ελλάδα μας δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ. Έχουμε 15 βουλευτές. Έχουμε 10 ακόμη δηλαδή, διότι 5 ήδη πήραν το λόγο. Κλείνουμε λοιπόν τώρα τον κατάλογο των ομιλητών. Δίνουμε το λόγο στον Ρομπέρτο Σοβαρία, μέλος του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Δύο λεπτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που με καλέσατε. Εγώ δεν θέλω... Ε, ε, εγώ δεν θέλω να... Να τσακωθώ με τον κύριο Ικούνεν σχετικά με τη Ρότα ε, σε Μεγάλη Κανάρια. Διότι χθε ήδη μας κατέφτασαν δεν ξέρω πόσοι μετανάστευσαν από αυτή τη Ρότα. Εμείς πάντοτε υποστηρίξαμε πολιτικές ε, συντονισμού, υποστηρίξαμε το Frontex και του συνοριακούς ελέγχους. Και η θέση μας διαφέρει από αυτήν του κυρίου Χούνκο. Αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι να βοηθήσουμε τον κύριο Μπουσουτήλ για να δει προς τα πού πάει το Frontex. Το Ισπανικό Κοινοβούλιο μίλησε ήδη για το, αποφάσισε ήδη για το θέμα της επικουρικότητας και σχετικά δηλαδή με τη δημιουργία εξ νόβο για, μια νέα οργάνωση, ε, για ένα νέο οργανισμό που θα ασχολείται με θέματα δικαιοσύνης και μετανάστευσης. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα θέμα απλούστευσης και λειτουργικότητας και σε μια περίοδο κρίσης θα έπρεπε να εφαρμόζουμε αυτές, αυτού του είδους τις αρχές δεν είναι ώρα να δημιουργούμε νέους οργανισμούς. Θέλουμε περισσότερο συντονισμό. Το καλύτερο λοιπόν θα ήταν η Frontex με μια μικροαλλαγή της διάρθρωσής της να αναλάβει τη διαχείριση αυτών των μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, να προχωρήσει στην διοικητική απλούστευση, στην εξοικονόμηση κτλ. Θα έχουμε δηλαδή μία αναλογικότητα των μέσων, θα μπορούσαμε δηλαδή να διευρύνουμε το πεδίο αρμοδιοτήτων της ε, Frontex, να την ενισχύσουμε. Οπότε η αναλογικότητα και η απλούστευση ως αρχές θα γινόταν σεβαστές. Θα ήθελα να ακούσω τι λέτε εσείς για την πρόταση που εμείς υποβάλαμε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Δύο λεπτά η κυρία Ματιού. Εγώ πιστεύω αντίθετα από ότι ο Γερμανός συνάδελφο ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης αφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Διότι όταν φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης μετά έρχονται όλοι, ε, ε, ε, διασκορπίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε στο Frontex. Όσοι εισηγήτρια στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πέρσι για τους οργανισμούς, πρέπει να σας πω ότι από πέρυσι φέτος διαπίστωσα ότι αυξήθηκε πολύ ο προϋπολογισμός σας μεν, αλλά δεν σας δόθηκαν τα μέσα διοικητικά κλπ για να μπορέσετε να ξοδέψετε αυτά τα λεφτά. Πρέπει λοιπόν να δείτε πώς θα ξοδέψετε αυτόν τον προϋπολογισμό διότι τα εξωτερικά μας σύνορα πρέπει να τα φυλάμε καλύτερα. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν είναι μόνο η ανθρώπινη απελπισία. Μέσα σε όλα αυτά κύριε Διευθυντά υπάρχουν όλα αυτά τα δίκτυα μαφίας και εγκληματικότητας τα οποία θα πρέπει να τα περιορίσουμε και με τον προϋπολογισμό που σας χορηγούμε και που ελέγχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουμε ότι να τα αξιοποιήσετε ούτως ώστε να καταπολεμήσετε όλα αυτά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δραβάρας, Ελληνικό Κοινοβούλιο, δύο λεπτά. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την εκδήλωση αυτή και την συζήτηση η οποία ξεκινάει για πολύ θεμελιώδη και πολύ σημαντικά θέματα. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι αποτελεί καταστατική σημασία στόχο της Ένωσης η δημιουργία του ενιαίου χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας αποτελεί το ίδιο καταστατικής σημασίας η πράξη, η δράση που έχει σχέση με τον καθορισμό των ορίων αυτού του χώρου. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για χώρο ενιαίο εάν δεν έχουμε φροντίσει να αναλάβουμε δράσεις για την προστασία αυτών των ορίων που στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτουν με τα εξωτερικά σύνορα αυτού του χώρου. επομένως αυτοί που ισχυρίζονται την κατάργηση της frontex προφανώς υιοθετούν αποδέχονται ή καλλιεργούν λογικές οι οποίες στρέφονται εναντίον αυτής της ίδιας της ευρωπαϊκής ένωσης αφού δεν μπορεί να νοηθεί διαφορετικά η καλλιεργουν λογικες οι οποιες τρεφονται εναντιον αυτης της ιδιας της ευρωπαικης ενωσης αφου δεν μπορει να νοηθει διαφορετικα η υπαρξη ενιαίου χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης χωρίς την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και βέβαια αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να συνοδεύεται με την αναγνώριση και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών των λαών οι οποίοι συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτά είναι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία απειλούνται από την παράνομη και την αθέμητη μετανάστευση αφού στο εσωτερικό των κρατών αυτών και κυρίως στο εσωτερικό της χώρας μου της ελλάδας και η εγκληματικότητα αυξάνεται και η ανασφάλεια καλλιεργείται. υπ' αυτή την έννοια θεωρώ απαράδεκτες θεωρώ αντιενωσιακές λογικές αυτές που προτείνουν την κατάργηση της frontex. αντιθέτως συμφωνώ με όσους μίλησαν για μια ανάπτυξη αυτού του οργανισμού για μια επέκταση των αρμοδιοτήτων του και κυρίως με την προσπάθεια που αποτελεί σύμφυτη και εγγενή με την αναγνώριση των δικαιωμάτων που έχουν σχέση με την προστασία του χώρου της ελευθερίας της δικαιοσύνης και της ασφάλειας και έχει να κάνει με την παροχή όλων των μέσων που είναι αναγκαία και απαραίτητα ώστε να είναι αποτελεσματική η φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Maritati, del Senato Italiano. Ο κύριος Μαρινάτη από την Ιταλική Γερουσία. Πολύ σύντομα. Η μετανάστευση είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Τι να πω εγώ μετά από αυτά που μας είπε ο Έλληνας συνάδελφος. Ε, είναι ευρωπαϊκό σύνορο και η Ιταλία. Τα Ιταλικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Πρέπει να έχουμε σαφή πολιτική για τη μετανάστευση. Πιστεύω λοιπόν ότι το Frontex θα πρέπει να αποτελεί ένα μέσο στην υπηρεσία όλων στην Ευρώπη. Να αποτελεί ένα μέσο για τον συντονισμό, τη γνώση και την υποστήριξη των κρατών, των αντίστοιχων κρατικών οργανισμών. Σε πολιτικό επίπεδο χρειάζεται να βρεθούν όμως λύσεις. Και αυτό γιατί, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα που μας ανέφερε ο συνάδελφος Γιούνκο όταν μιλούσε για στρατόπεδα, για λάγκερ και η Ιταλία θα πρέπει να προσέχει πριν αρχίσει να υπογράφει συμφωνίες σαν αυτές που υπέγραψε με τη Λιβύη που οδήγησε στη δημιουργία στρατόπεδων συγκέντρωσης δίνοντας ε, χρήματα στη Λιβύη, τα οποία πώς χρησιμοποιούνται μετά. Τα λιβικά, οι λιβικές ε, περιπολίες πυροβολούν τα δικά μας ψαροκάικα. Αν εμείς λοιπόν θέλουμε να είμαστε φάρος πολιτισμού, πρέπει να κοιτάξουμε να δρούμε διαφορετικά για να μην γίνουμε ένας πόλος πολιτιστικής οπισθοχώρησης. Η κυρία Ρομέρο Λόπες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Και εγώ Ισπανίδα είμαι. Και ήμουν εθνική βουλευτής όταν πιέσαμε από την νότια η Ισπανία για να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός που θα έδινε προστιθέμενη αξία στα δρόμενα της Ευρώπης για τις ευαίσθητες περιοχές όπως η Νότια Ισπανία και τα Κανάρια νησιά. Είχαμε φανταστεί αυτόν τον οργανισμό ως έναν οργανισμό για την αποφυγή τραγωδιών και ναυαγίων. Διότι Στα Σαπιοκάραβα τι γινότανε. Ερχότανε Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν κατάλαβα τι συνέβη με το κινητό μου, λέει η ομιλήτρια για τους μικροφωνισμούς. Θελήσαμε λοιπόν να αποφύγουμε με τη Frontex τη δημιουργία τραγωδιών, να αποφύγουμε μαζί με τα σαπιοκάραβα πέρα από τους μετανάστες να έρχονται και εγκληματίες. Αλλά τι έγινε. Συνδέσαμε εμείς τη Frontex με την Europol. Άλλο πράγμα είναι η οι, οι έμποροι ναρκωτικών, άλλο οι σωματέμποροι, άλλο οι φουκαράδες μετανάστες που έρχονται με τα πλοιάρια. Πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα να γίνονται χωριστά. Πρέπει να ξεχωρίζουμε ε, δεν θα μπορέσουμε εμείς να ξεχωρίζουμε πραγματικά αυτούς που είναι οι αιτούντες άσυλο δεν θα μπορέσουμε αυτού, να αντιμετωπίσουμε με ανθρώπινους όρους αυτούς τους παράνομους οι οποίοι έρχονται όντως όμως για δουλειά και δεν θα μπορούμε, να τους ξεχωρίζουμε όλους αυτούς με τους ε, εγκληματίες. Λοιπόν, γιατί η Europol δεν αφήνει ήσυχου τους, ε, τους ε, λαθρομετανάστες και δεν ψάχνει να βρει τους σωματέμπορους και τους διακινητές των μεταναστών, δεν θα έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο. Ο κύριος Χάιντς Μάουρους από το Bundesrat Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συναντηθούμε και να συζητήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους κυρίους Λαϊτίνεν και Πουσοτήλ για τις παρουσιάσεις τους. Ε, ζήτησα όμως το λόγο ε, για να απαντήσω στον συνάδελφο Χούγκο. και μιλώ και στο όνομα του συναδέλφου Πέρενς από το ε, Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Η θέση του κυρίου Χούγκο είναι η θέση η δική του και του, της, και του κόμματός του, όχι του ε, Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Όσον αφορά το θέμα της λαθρομετανάστευσης και την αύξηση της, ε, του οργανωμένου εγκλήματος, ε, είναι απαραίτητο να αντιδράσουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται μια συνεργασία η οποία μπορεί να ε, βελτιωθεί συνεργασία ανάμεσα στη Frontex ε, και στις αρχές που είναι υπεύθυνε για την ε, ε, αντιμετώπιση της εγκληματικότητα. Εγώ θα ήθελα ενίσχυση της Frontex, η αντίδραση αυτή είναι απαραίτητη στο δεδομένο των εξελίξεων. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέ για όλους μας. Ευχαριστώ κυρία Βερζάτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ιούνκο, τον οποίο συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις του για το ρόλο της Frontex που σήμερα συμπεριφέρεται για να μην μπούμε, να μην φτάσουμε ως εκεί, ως ένα όργανο κλεισίματος των συνόρων. Θα ήθελα τα λίγα καλά στα οποία συνεισφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας να εφαρμοστούν προσχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Δύο εκθέσεις έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι η συγγήτρα των δύο αυτών εκθέσεων και θα ξεψηρίσουμε πραγματικά τους όρους με τους οποίους γίνεται ασκείται μάλλον η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Και εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου τις απόψεις με την, για τη συμφωνία με τη Λιβύη, όπως και αυτή της Τινησίας δηλαδή. Πρόκειται για ατιμωτικές συμφωνίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εδώ δεν είναι μόνο το να σεβαστούμε ένα ελάχιστο ευζοίας και ευημερίας για αυτούς τους ανθρώπους που επαναπατρίζουμε. Πρόκειται για την εφαρμογή τη Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε εμείς ε, να τους στέλνουμε πίσω σαν ανσακιά. Και ναι, εμείς προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, αλλά θα πρέπει να δίνουμε και το καλό παράδειγμα εμείς ήδη για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η μεταναστευτική πολιτική είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι λύση τη στιγμή της παγκοσμιοποίησης. Άμα δείτε και τα δημογραφικά προβλήματα τα οποία έχουμε, δεν είναι ώρα να κλείνουμε τις πόρτες. Ο κύριος Σταβάρες. Τα πιο πολλά ήδη έχουν υποθεί. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μία αφορά στην ανθρωπιστική πλευρά αυτών των αδαγίων σαρέματος ε, των ε, μεταναστών σε ανοιχτή θάλασσα, μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο κλπ. Πριν από λίγο καιρό, συζητήθηκε ένα θέμα που αφορά όλες αυτές τις επιχειρήσεις ανοιχτής θάλασσας. Και τίθεται το θέμα σε σχέση με αυτά εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να εγκριθεί το περιεχόμενο και να υλοποιηθεί η πρακτική πάντα σε σχέση με, με την κατεύθυνση να υπάρχει διάσωση ζωής ε, στην ανοιχτή θάλασσα και να δράσουμε σε σχέση με ανθρωπιστικές σκέψεις και να διασφαλίσουμε ότι η αρχή της ε, μη απέλασης ε, θα εφαρμόζεται. Δεύτερον, η σχέση, η ερώτηση για τη Λιβύα δεν ε, μπορεί, δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζεται ο σεβασμό για τα δικαιώματα των μεταναστών και εκείνων που ετούνται άσυλο. Το να παραδίδονται σε μια χώρα που δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τα δικαιώματά τους είναι μια έμεση παραβίαση όσον αφορά τη σύμβαση της ε, Γενέβη. Ε, ή σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με γεγονότα όπως ε, την επίθεση κατά των Ιταλών αλλιέων. Και πρέπει εδώ να το δούμε αυτό. Σε οποιαδήποτε κατάσταση ε, τέτοιας αντιμετώπισης ή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα με τη Λιβύη ή διαφορετικά θα ανοίξουν οι πύλες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία τοποθέτηση και βεβαίωση για να συνεισφέρουμε στη συζήτηση. Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμοδιότητα αποκλειστική, αποκλειστική των κρατών μελών και όχι της Frontex. Εντάξει, λοιπόν τι κάνει και τι είναι η Frontex. Είναι συντονιστικός ρόλος, συνεργασία, είναι ανάλυση στρατηγικών στοιχείων, είναι οι επιστροφές, από κοινού επανεισδοχές ή απελάσεις συνεργαζόμαστε ώστε και στο υπόλοιπο να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι δεν έχει καμιά αρμοδιότητα η Frontex για την, τον διοικητικό χαρακτήρα των κέντρων υποδοχή. Είναι θέματα που πρέπει να αποσαφινιστούν πλήρω για να μην υπάρχουν παρανοήσει. Και τώρα για τον Σάιμον Μπούσουτιλ και, την ερώτηση, μια, και τη συζήτηση. Μια ερώτηση. Σε στιγμέ κρίση πίεσης μεταναστευτικής, ένα συγκεκριμένο σημείο των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να υποχρεώσουμε κάποιον να εκφράσει αλληλεγγύη. Δεν είναι επουσιώδες αυτό το ερώτημα, είναι σημαντικό. Μπορεί να είναι υποχρεωτική η έκφραση αλληλεγγύης σε μια κρίσιμη στιγμή πίεσης μεταναστευτικής. Ε, σε αυτό το ερώτημα πρέπει να δοθεί απάντηση. Και δεύτερον, που συσχετίζεται ω ερώτημα με το πρώτο. Κύριε Διευθυντά, κύριε Λάιτίνεν, ποιος είναι ο βαθμός ε, δέσμευσης ε, όσον αφορά την τον κατάλογο των μέσων που διατίθενται από πλευράς της Frontex για να αντιμετωπιστούν προσωρινά, να αντιμετωπιστεί μια κρίση μεταναστευτική πίεση σε ένα συγκεκριμένο ή σε κάποια συγκεκριμένα μεθοριακά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ε, σας παρακαλούμε τώρα εσά να είσαστε παρακαλώ, σύντομοι στην παρέμβασή σα. Okay, ευχαριστώ και ελπίζω ότι ο Διευθυντής Λάιτινεν θα είναι σε θέση να απαντήσει για κάποια από αυτά τα σημεία, διότι δεν ακούστηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις. Θέλω να σκεφτούμε αυτούς που αποβίωσαν στη Μεσόγειο και τι γίνεται σε σχέση με τις ε, ε περιπολίες που πολλές φορές σε σχέση με τρίτες χώρες όπως την Λιβύη επαφίενται. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό και από πλευράς του συναδέφου Ρούι Ταβάρες για το γεγονός το οποίο ανέφερε για την ύπαρξη αυτών των ε, δυνατοτήτων όμως ε, η Λιβύη ε, πετέθη σε Ιταλούς αλληλείς από πλευράς τους. Δεν ήταν μόνο απειλή, πυροβόλησαν κατά των ατόμων αυτών των Ιταλών αλληλείων Τι πιστεύετε λοιπόν εσείς γι' αυτό, για τέτοια γεγονότα, για αυτό το οποίο συμβαίνουν, για αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά την αποβίβαση για παράδειγμα 100 150 μεταναστών σήμερα που αποβιβάστηκαν και κάποιον χάθηκαν τα ίχνη. Ίσως έχουν αποβιώσει αυτοί οι άνθρωποι. Τι συμβαίνει λοιπόν. Ίσως τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να μην υποτιμούμε, να μην υποβαθμίζουμε την εμβέλεια αυτών των ε, ζητημάτων. Θέλω να εκφράσω τις ε, ευχαριστίες μου για αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Πρέπει να είμαστε πράγματι σε γρήγορση, να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τον δημοκρατικό έλεγχο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατιωτικέ περιπολίε. Σα ευχαριστώ, έχουμε ήδη καθυστερήσει και παρακαλώ σε αυτόν τον τελευταίο γύρο για να κλείσει αυτή η πρώτη συνάντηση εργασία μα να είσαστε το δυνατό δυνατόν συντομότερο. Ξεκινώντας πρώτα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Frontex, κύριο Λάτινεν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ φυσικά πολύ για όλους τους ε, όσους συμμετείχαν σε αυτή τη ζωντανή συζήτηση. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα και λόγω πίεσης χρόνου όλα τα ερωτήματα δεν μπορώ να τα απαντήσω αλλά επικεντρωνόμενο στη συζήτηση στα ουσιοδέστερα θέματα θα ήθελα να τοποθετηθώ επ' αυτών. Πρώτο σημείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ευθύνη του ελέγχου των συνόρων είναι ευθύνη των κρατών μελών. Η Frontex <clears throat> δεν έχει κανένα, καμιά εκτελεστική αρμοδιότητα, οποιαδήποτε εκτελεστική αρμοδιότητα δεν υπάρχει από πλευρά τη Frontex. Όλε οι αποφάσει λαμβάνονται από τα όργανα και του φορεί των κρατών μελών και του δικού του συνοριοφύλακε. Εμεί κάνουμε μια ανάλυση κινδύνου. Δίνουμε στα κράτη-μέλη αυτά τα στοιχεία για από κοινού συντονισμό και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρηματοδοτούμενε εν μέρη με αυτόν τον τρόπο και προσπαθώντα να προαγάγουμε, να προαχθεί η ικανότητα των συνορεφυλάκων των κρατών μελών να ακολουθήσουν τους κανόνες, τις πολιτικές και την ομοθεσία του, της, των, Ευρωπα, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όταν έρχεται το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ουσιώδες σε αυτό, θα ήθελα να υπενθυμίσω το πρώτο σε πρώτο επίπεδο ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι αρμόδιος για την λήψη αποφάσεων. Δεν είναι η Frontex. Είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που λαμβάνουν αποφάσεις για την εισδοχή κάποιων ατόμων ή για την μη εισδοχή τους. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι το, της Frontex. Αν το θέσουμε σε λειτουργική κλίμακα, σε συνεργασία, αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη, από τους ίδιους και ποιο είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας ε, από την Frontex, 11.000 ε, <clears throat> επιχειρήσεις ε, γίνονται ετήσια με ένα προϋπολογισμό λιγότερο από 90 εκατομμύρια ευρώ έχουμε 270 στελέχη. Συλλέγουμε περίπου 2.000 συνοριοφύλακε που δρούν σε αυτά τα πλαίσια. Τα κράτη-μέλη έχουν 400.000 συνοριοφύλακε και δεν είμαι καν σε θέση να πω ποιο είναι ο συνολικός προπολογισμό που δίνουν κονδύ, ως κονδύλια τα κράτη-μέλη στους συνοριοφύλακες τους. Μία πτυχή την οποία δεν έχουμε συζητήσει εδώ ακόμα είναι το capacity building aspect, η πτυχή της δυνατότητας ανάπτυξης του δυναμικού. Είπε ο κ. Μπουσούτιλ ότι έχουμε ένα κοινό ε, στόχο και ένα κοινό, ας το πω έτσι, πρότυπο που έχει συνταχθεί από τα κράτη-μέλη αλλά και τους ε, ε, εταίρους μας, την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες για παράδειγμα, που έχει συνεισφέρει σε αυτό το curriculum, σε, αυτή την ατζέντα, το θεματολόγιο για τους πρόσφυγες. Η, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι, ας το πω έτσι, θεμελιώδης προσέγγιση της Ευρώπης για τα θέματα ελέγχου των συνόρων ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με του νεοφύλακε των κρατών μελών, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, σε κοινέ δράσει, σε οτιδήποτε είναι δυνατόν να κάνουμε, λαμβάνουμε ιδιαίτερη μέρη να προσέξουμε και για του δικού μα ε, τα δικά μα στελέχη, με την κατάρτιση και την εκπαίδευση, να διευρυνθούν οι γνώσει του. Είχαμε μια εξαιρετική, ε, α το πω έτσι, ημερίδα κατά θεμελιώδει δικαιώματα και αυτή ή περίοδο κατάρτιση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτή η συνεργασία προ αυτή την κατεύθυνση συνεχίζεται. Και όταν έχουμε την εξέταση και σε σχέση με τρίτε χώρε που είναι εταίροι μα, το θέμα είναι θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε με του εταίρου μα ε, των τρίτων χωρών ε, για να προαχθεί ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η καλύτερη οδό είναι να του απομονώσουμε και να μην λαμβάνονται αυτέ οι πτυχέ υπόψη από πλευρά του ή να μην λαμβάνονται τέτοιου είδου πρωτοβουλίε καν. Αυτό που θα ήθελα να πω όμω εν κατακλείδη είναι βλέπουμε να εμένουν οι περιπτώσεις τραγωδιών στην, στην ανοιχτή θάλασσα. Ποιος είναι ο πρώτος και κύριος ρόλος των λιμενοφύλακων και των λιμενικών αρχών. Πιστέψε με, είναι το να διασώζονται ανθρώπινες ζωές. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, πολύ δύσκολη δουλειά και σε όλα αυτά τα συμβάντα που συμβαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα για την ε, αναζήτηση και διάσωση στην ανοιχτή θάλασσα, αυτός είναι ο πρώτος και κύριος ε, λόγος και ρόλος. Διάσωση των ανθρώπων ανθρώπων. Αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω και να τονίσω για άλλη μια φορά σε σχέση με την αξιολόγηση του δυναμικού και των δυνατοτήτων των κρατών μελών. Μέχρι στιγμής δεν είναι αυτός ο ρόλος ε, της Frontex. Δεν δίνουμε δηλώσεις ή τοποθετήσεις σε σχέση με τις αρμοδιότητες και το δυναμικό και τις ικανότητες των επιμέρους κρατών μελών. Γι' αυτό το σκοπό υπάρχουν θεσμικά όργανα και μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπως όμως είπα στην δική μου εισαγωγή, η καταπολέμηση του εγκλήματος στα εξωτερικά σύνορα είναι κάτι καινούριο σε ευκαιρία. Ο κύριος Κούκελμπεργκ ανέφερε τον μηχανισμό συντονισμού και με ιδιαίτερη χαρά βλέπω τον συνάδελφο από την Europol που σύντομα θα παρέμβει και βλέπουμε ότι σε καθημερινή βάση υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο θεσμικών οργάνων Frontex και Europol. Καθορίζουμε φυσικά τον ρόλο μας, τον ρόλο μας για τις ξεχωριστές μας δράσεις, δράσεις Frontex και δράσεις Europol. Καθημερινή συνεργασία με σαφείς διαχωριστικές γραμμές. Δυστυχώς δεν έχω την ευκαιρία ευκαιρία να απαντήσω αναερώτηση και ερώτημα. Αλλά υπάρχει ανάγκη να, σε περίπτωση ύπαρξη ανάγκη να επικεντρωθώ σε κάποιε ε, από αυτέ τι ερωτήσει, θα υποβάλω τι απαντήσει γραπτό. Ο χρόνο πιέζει. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Κατανοείτε και σα ευχαριστούμε γι' αυτό του περιορισμού του χρόνου. Και σε σχέση με τις εισαγωγικέ ε, παρατηρήσεις, εσείς κύριε από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα θέλετε να απαντήσετε όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Και στην εισαγωγική μου παρέμβαση είπα ότι θα αναφερθώ στις επικρίσεις κάποιων οργανώσεων ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει και μία νομική γνωμοδότηση του 2007 της Προαζήλ και της, ε, Amnesty, και της Διεθνούς Αμνηστίας. Το αποτέλεσμα ε, εκφράζεται ως εξής, ε, ότι η Ευρώπη απομονώνεται από πρόσφυγες και μετανάστες και ότι το σχέδιο αυτό ε, δεν σέβεται τα, τις ε, νομικές και άλλες υποχρεώσεις ε, των κρατών μελών. Φυσικά είναι αλήθεια ότι η Frontex δεν εφαρμόζει όλα τα μέτρα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το ερώτημα είναι προς τα που εξελίσσεται, προς ποια κατεύθυνση εξελίσσεται το καθεστώς συνόρων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κεντρικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό οι επικρίσεις όσον αφορά τις εξελίξεις αυτές είναι πολύ σημαντικέ, διότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική πτυχή τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ε, και τέλο, για να κλείσουμε το πρώτο αυτό μέρο, ο κύριο Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να απαντήσω στην ε, παρέμβαση του κυρίου Χούγκο όπου, ότι η Frontex ε, ελέγχει τους πρόσφυγε. Όχι, δεν έχει τον έλεγχο και είναι σημαντικό να γίνει διάκριση ανάμεσα στις αρμοδιότητες στα εξωτερικά σύνορα και τις αρμοδιότητες για θέματα που έχουν να κάνουν με το άσυλο. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια νέα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ε, υπηρεσία στήριξης ε, για την υποβολή της ονασύλου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τους πρόσφυγες σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ο κύριος Καλαζεύσκη ρώτησε εάν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για μια υπερ-υπηρεσία ή για μια δευτερεύουσα υπηρεσία, μια βοηθητική. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία από τις ε, ε, τροπολογίες που προτείνονται έχει να κάνει με την δυνατότητα της Frontex να αγοράζει ή να νοικιάζει τον δικό της εξοπλισμό. Εάν γίνει αυτό, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί ο προπολογισμό της Frontex. Τρίτον, ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κατανοητό ότι πολλοί κόσμος έχει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στη Βαρσοβία με αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το θέμα αυτό βρισκόταν στην κορυφή της ημερησία ημερήσιας διάταξής μας. Ρώτησα πολλά πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μαντέψτε, μας απαντήσανε σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλά νομίζω ότι η πιο σημαντική απάντηση που λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, Βαρσοβία ήταν ότι η ε, Frontex μας είπε πολύ σαφώς ότι έχει μηδενική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν έστω και ένας ε, συνοριοφύλακας που συμμετέχει στις επιχειρήσεις παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν θα συνδέεται πια με τη Frontex. Μία υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και αυτό πάντα θα αναφέρεται στην έκθεσή μου. Τέταρτον, η δημιουργία της νέας υπηρεσίας πληροφορικής που ανέφερε ο κύριος Σοραβία από την Ισπανία. Ο κύριος Σοραβία δεν συμφωνεί με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών. Αυτό θα πρέπει να το μεταφέρω στον συνάδελφό μου, τον κύριο Κάρλος Κοέγιο. Ο κύριος Σοραβία λέει ότι η, η λειτουργία αυτή θα πρέπει ε, να ε, δοθεί στην Frontex. Η νέα υπηρεσία όμω, πιθανότατα να αναφερθεί αύριο ε, κατά το τμήμα τη συζήτηση που έχει να κάνει με το Σέγγεν. Ε, Επίση, μου άρεσε πολύ η παρέμβαση του κυρίου Τζαβάρα από την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα μέσα για να λειτουργήσουν όλα αυτά. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτή η δήλωση προέρχεται από κάποιον από την Ελλάδα, που τυχαίνει να είναι η χώρα που αντιμετωπίζει τι χειρότερε δυσκολίε όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε το εξή, και είναι πολύ σαφέ αυτό. Η Frontex επιφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απάντησή μου είναι ότι η Frontex μπορεί να επιφέρει προστιθέμενη αξία. Λέω ότι μπορεί και όχι ότι επιφέρει, διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά από αυτή που κάνει μέχρι τώρα. Επίσης ε, αναφέρθηκε το θέμα των αρμοδιοτήτων. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η συνθήκη καθιστά απόλυτα σαφές ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι ε, αρμοδιότητα των κυριάρχων κρατών. Υπάρχει όμως ένα αλλά πολύ σημαντικό. Το άρθρο 2ε του κανονισμού Frontex ε, και το διαβάζω λέει σαφώς ότι η Frontex θα πρέπει επίσης να έχει ω καθήκον να βοηθάει τα κράτη-μέλη υπό συνθήκε που απαιτούν αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια στα εξωτερικά σύνορα. Ναι, κάθε κράτο είναι κυρίαρχο, αλλά όταν ένα κράτο αντιμετωπίζει δυσκολίε, θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή που με φέρνει στο τελικό μου συμπέρασμα. Την αλληλεγγύη που πολύ σωστά έθιξε ο κύριο Δία Δεμέρα. Ναι, πρέπει να επιδιώξουμε την αλληλεγγύη και θα πρέπει να επιδιώξουμε μια αλληλεγγύη λειτουργική. Τώρα, είτε αυτή είναι προαιρετική είτε είναι υποχρεωτική αλληλεγγύη, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Σημαντικό είναι να λειτουργεί. Μέχρι στιγμή δεν έχει λειτουργήσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάθε προσπάθεια για να λειτουργήσει καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποσούτιλ, ευχαριστώ κύριε Χούγκο, ευχαριστώ κύριε Λαϊτίνεν, ευχαριστώ και όλου του βουλευτέ που πήραν το λόγο. Ήταν μια ιδιαίτερα επικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαστε πεπισμένοι ότι η δεύτερη συζήτηση που θα ξεκινήσει τώρα δεν θα είναι ε, λιγότερο ενδιαφέρουσα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν ε, το πάνελ της πρώτης συζήτησης και χωρίς διακοπή για να προλάβουμε, διότι μία ώρα μας απομένει. Σας παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι μας πιέζει ο χρόνος ε, των διερμηνέων, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ λοιπόν χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσουμε στη δεύτερη συζήτηση. Καλώ τον κύριο Ρομπ Βέινράιτ, που είναι διευθυντής της ε, Europol, τον κύριο Αωτίντια Φεβέρα, που είναι μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ υπεύθυνο για την έκθεση της Europol και τον Λόρδο Πίτερ Μπάουνες που είναι πρόεδρος της Υπό Επιτροπή Δικαιοσύνη και Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Thank Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία σας. διότι η δεύτερη αυτή συζήτηση είναι υψής της σημασίας και συνδέεται με την Europol. Μία ώρα έχουμε μπροστά μας. Σας παρακαλώ. Οι εισαγωγικέ παρεμβάσεις των τριών ομιλητών να διαρκέσουν λιγότερο από 10 λεπτά, ώστε να δώσουμε το πολύ δύο λεπτά στους βουλευτές που θα θέλουν να παρέμβουν μετά. Προχωράμε λοιπόν κατευθείαν. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρομπ Βέινραιτ, που είναι διευθυντής της Europol. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές, σας ευχαριστώ που με καλέσατε στη σημερινή συζήτηση και που μου δίνετε τη τιμή να ανοίξω τη σημαντική αυτή συζήτηση για την Europol. Το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσία της Europol έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια και θα έχουμε ακόμα κάποιες τα επόμενα χρόνια. Θα αναφερθώ σε αυτές στην παρέμβασή μου. Θα ήθελα όμως επίσης να ε, σας παρουσιάσω το έργο της Europol ώστε να έχουμε ένα καλό πλαίσιο για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ε, η Europol είναι η υπηρεσία επιβολής του νόμου. Δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τους πολίτες της Ευρώπης, να ε, προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθώντας τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν την απειλή του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Την ε, υπηρεσία μας τη δημιουργούμε με έναν τρόπο που θεωρώ ότι αποτελεί συντονισμένη ε, ανταπόκριση απέναντι στις ε, πιο σημαντικέ απειλέ που ε, αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Το κάνουμε αυτό διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. 650 εμπειρογνώμονες, αναλυτές και αξιωματικούς επιβολής του νόμου απασχολούμε από τις από τα κράτη-μέλη με προϋπολογισμό περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη βασίζονται στις υπηρεσίες μας 24 ώρες το 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα για να συντονίσουν περίπου 14.000 διασυνοριακές επιχειρήσεις το χρόνο εν μέρη κατά κάποιον από τις, τα πιο ε, επικίνδυνα δίκτυα που λειτουργούν στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητε αυτές έχουν οδηγήσει σε πολλές ε, συλλήψεις ε, και σε ε, διάσωση πολλών ε, θυμάτων, ε, μεταξύ άλλων παιδιών καθώς και στην επιστροφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ από κέρδη του εγκλήματος. Ένα παράδειγμα της δουλειάς μας από τις 14.000 αυτές επιχειρήσεις το χρόνο είναι μια πρόσφατη επιχείρηση για ανθρώπους που κακοποιούν ανήλικους στο ίντερνετ. 225 ε, ανθρώπους εντοπίσαμε, οι 115 έχουν ε, ε, συλληφθεί. Οι έρευνές μας πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε 19 χώρες ώστε να δώσουμε τέλος στο φοβερό αυτό έγκλημα το οποίο διαπράτεται μέσω του διαδικτύου. Και πρόκειται για τυπική περίπτωση του πώς η Europol μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλύσει πολύπλοκα εγκληματικά στοιχεία, να εντοπίσει εγκληματικά δίκτυα και να χρησιμοποιήσει τις ε, υπηρεσίες ε, πλατφόρμας ε, για να συντονίσει τις δραστηριότητες, τις αναλύσεις, να τις μετατρέψει σε αποτελεσματική αστυνομική δράση ε, στην πράξη ώστε να αποτρέψει ε, περαιτέρω ε, βλάβη στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η Europol δεν μπορεί να αναγκάσει κανένα να κάνει κάτι. Βασιζόμαστε στην συνεργασία των κρατών μελών για την ε, ανάπτυξη του αστυνομικού δυναμικού μας ε, και λειτουργούμε ως κέντρο πληροφοριών για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα της Europol να παρέχει υπηρεσίες πλατφόρμας μέσω των οποίων οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ευρώπη να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Μας ενδιαφέρει η προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων ε, είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό για τους πολίτες μας και τα κοινοβούλια μας. Ε, πιο σημαντικό όμως είναι ότι η δουλειά της Europol είναι να κάνει την Ευρώπη πιο ασφαλή προστατεύοντας τους πολίτες μας από το διεθνές έγκλημα και την τρομοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική για μας η κατανόηση του κοινού και γι' αυτό επικροτούμε κάθε ε, προσπάθεια να βελτιωθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία. Η ε, θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχει επιφέρει πολλέ ε, αλλαγέ στη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στον τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών. Και όσον αφορά την λογοδοσία, έχουν γίνει κάποιες σημαντικές βελτιώσεις. Η Europol, ωστόσο, έχει διαφορετική ιστορία σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Δημιουργηθήκαμε πριν 10 χρόνια με βάση ε, διακυβερνητικές ρυθμίσεις ε, που τότε, ε, ενεργώντας υπό τον τρίτο πυλώνα τότε, θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική εμπλοκή στη δουλειά μας ήταν περιορισμένη τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εμπλέκονταν ε, άμεσα και το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, το μοιράζονταν η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ε, Συμβούλιο λοιπόν ήταν ο θεματοφύλακας των εθνικών συμφερόντων και των Ευρωπαίων πολιτών. Μέχρι τη φετινή χρονιά η Europol ήταν, λογοδοτούσε στο Συμβούλιο Υπουργών και στο διαχειριστικό της Συμβούλιο με την ε, επικύρωση της ε, σύμβασης ε, Europol και, τα σχετικά, και των σχετικών πρωτοκόλων εμπλέκονταν τα, οι εθνικές κυβερνήσεις. Όπως σας είπα, λοιπόν, επικροτούμε τις τροποποίησεις που έχουν γίνει. Πιστεύω ότι η θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λιζαβόνας ήταν σημαντική βελτίωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν ιδιαίτερα καλή ευκαιρία για μα να αυξήσουμε την διαφάνεια εντός τη Europol. Η συνθήκη ε, θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια στην καρδιά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δημιουργεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για την Europol και νέο πλαίσιο για δημοκρατική λογοδοσία. Σύμφωνα με τι νέε ρυθμίσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η Europol ε, συνεχίζει να ε, είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί στο διαχειριστικό τη Συμβούλιο, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κάθε νέα νομοθετική πράξη στον τομέα αυτόν υιοθετείται με την διαδικασία της ε, συναπόφασης. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα συμμετέχει από την αρχή στη διαδικασία αυτή και θα έχει και δικαίωμα αρνησικυρίας. Τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, λαμβάνουν ε, διάφορα έγγραφα από το Europol και επίσης θα συμμετέχουν στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης ε, των ε, δράσεων στον ε, τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών. Τέλος, ένας μελλοντικό κανονισμός Europol θα ρυθμίζει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Europol από το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα θα το συμβουλευόμαστε για θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή συνεργασία. Πέρα από την νέα συνθήκη της Λισαβόνας, η νέα βάση της Europol ενισχύει και τον μηχανισμό δημοκρατικής λογοδοσίας, ε, βελτιώνει επίσης την, ε, τις επιχειρήσεις μας, διότι μας βοηθάει να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην ε, καρδιά της νέας αρχιτεκτονικής για την εσωτερική ασφάλεια και προωθεί την πιο αποτελεσματική συνεργασία με την Frontex και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Με βάση την ανάπτυξη των δικών μας ρόλων, ε, προσβλέπω στην ε, αυξημένη συνεργασία της Europol με τη Frontex και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, ο ε, έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύεται ώστε να διασφαλιστεί η λογοδοσία της Europol. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η αρχή προπολογισμού της Europol ε, συνυπεύθυνη μαζί με το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν ε, το Κοινοβούλιο να χορηγεί απαλλαγή στον Διευθύντη όσον αφορά την, εφαρμογή του προϋπολογισμού, την εκτέλεση του προπολογισμού. Μπορεί επίσης ε, να απαιτεί απαντήσεις για θέματα και θα λαμβάνει και έκθεση από τον, έκθεση από τον Διευθυντή της Europol. Αυτά είναι πρακτικά μέτρα τα οποία με τα επιτρέπουν σε πράξη τι ρυθμίσεις για την ε, λογοδοσία της Europol. Ε, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της προστασίας δεδομένων, πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και για τους πολίτες. Αναγνωρίζω ότι η Europol έχει μοναδικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό να συλλέγει και να ε, αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να στηρίξουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Είμαι όμως και περήφανος που μπορώ να πω ότι η Europol το κάνει αυτό εντός ε, ενός πολύ ισχυρού πλαισίου ε, προστασίας των δεδομένων. Είναι μοναδικό στον κόσμο, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 15 χρόνια και πιστεύω ότι πετυχαίνει την ε, σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν περιορίζεται σε θέματα προϋπολογισμού. Η ε, εφαρμογή της ε, απόφασης του Συμβουλίου ε, έχει αυξήσει την λογοδοσία μας προς το Κοινοβούλιο με την υποβολή ετησίων εκθέσεων και το Κοινοβούλιο μπορεί να, ζητήσει, να καλέσει τον Διευθυντή για να συζητήσει θέματα που σχετίζονται με την Europol. Τέλος, κάθε τέσσερα χρόνια το Διευθυντικό Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέτει την διαξαγωγή εξωτερικής ανεξάρτητης έκθεσης για τις δραστηριότητε της Europol. Κοιτώντας το μέλλον και τον ε, προβλεπόμενο κανονισμό Europol. Η απόφαση του Συμβουλίου ήδη θέτει το πλαίσιο. Η Κομισιόν όμως θα προτείνει νέα νομική βάση για την Europol με βάση το άρθρο 88 της ε, συνθήκης και πιστεύω ότι αυτό ε, αποτελεί ε, νέα ευκαιρία να βελτιώσουμε τις ρυθμίσεις μας περί υποχρέωσης λογοδοσίας. Είναι επίσης τρόπος το η Europol να στηρίξει τις ε, εθνικές αστυνομικέ υπηρεσίε στην καταπολέμηση του εγκλήματο. Η Επίτροπο Μάνστρομ έχει προτείνει οδικό χάρτη για την τροποποίηση τη νομική βάση τη Europol που ε, συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση τη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου μας ε, του φετινού. αυτό είναι σημαντικό διότι η Europol ήδη έχει δαπανίσει πολύ χρόνο και ενέργεια για να προσαρμοστεί στο νέο νομικό πλαίσιο και πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ε, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αποτελεσματικό κανονισμό για τη Europol μαζί με την Κομισιόν ε, και ε, εκπροσώπους της Επιτροπής Λίμπη, ιδιαίτερα τον κύριο Διεθεμέρα, τους εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων και εκπροσώπους ε, του Διευθυντικού Συμβουλίου της Europol έχουμε εξετάσει πώς μπορούμε να κάνουμε τις ε, σωστές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση αυτή που θα αποτελεί το πρώτο στάδιο στον οδικό χάρτη προς ε, ένα νέο κανονισμό της Europol. Αυτή είναι πολύ σημαντική διαδικασία, μάλλον είναι η τελευταία μεγάλη αναδιοργάνωση εντός της Europol για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάτι χρήσιμο, όχι μόνο όσον αφορά τις ρυθμίσεις ε, δημοκρατικής λογοδοσίας αλλά και όσον αφορά την ε, ικανότητα της ε, κεντρικής αστυνομικής υπηρεσίας για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε την εντολή μας, ιδιαίτερα στους τομείς διασυνοριακού εγκλήματος, όπου είναι όλο και πιο δύσκολο να καταπολεμηθεί σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα όσον αφορά το κυβέρνο έγκλημα, την ομιμοποίηση παράνομων εσόδων και την ε, μεταφορά ε, κεφαλαίων ε, σε κλιματικές οργανώσεις. Επικροτούμε λοιπόν την ενίσχυση των, της υποχρέωσης λογοδοσίας της, Europol απέναντι στο εθνικό και, στα εθνικά και στο Ευρωκοινοβούλιο, την βελτίωση της συνεργασίας με τη Frontex και την αύξηση της δυνατότητας της Europol να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Κύριε Δίας Δεμέρα, δέκα λεπτά τουλάχιστον για την παρουσίασή σας. Χαίρετο με ιδιαίτερη συμπάθεια το Διευθυντή της Ευρωπόλ και τον συνάδελφο από τη Βουλή του Λόρδων. Χαιρετώ επίσης όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια με ιδιαίτερη συμπάθεια τους συναδέλφους από το δικό μου κοινοβούλιο, από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Τώρα να σας πω κάτι πολύ ειλικρινές. Εγώ ψάχνω, τη, αναζητώ τη διαθεσμική συνεργασία. Όλοι σας περιμένετε και αναρωτιέστε μα τι θα μας πει αυτός. Εγώ θα κοιτάξω να σας πω κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ με την πραγματικότητα. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε ο Διευθυντής. Αλλά αυτό το κοινοβούλιο δεν είχε την τόσο την αντίστοιχη ευτυχή ιστορία σε νομοθετικό επίπεδο. Η Σύμβαση Ευρωπόλ και τα τρία πρωτόκολλα προχωρούσαν πολύ πιο αργά από ό,τι προχωρούσε το οργανωμένο έγκλημα και το, η συνθήκη του Άμστερνταμ βρήκε την νομική μόρφη, τη νομική, έδωσε την νομική δυνατότητα για τη λύση του προβλήματος. Βρεθήκαμε λοιπόν εμείς σε παγίδα, δηλαδή στη νομοθετική, στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αποφάσισε το Συμβούλιο Ερήμην. Και ακόμη έτσι λειτουργεί η Europol. Πρέπει λοιπόν το σώμα να ξέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο του Συμβουλίου με 62 τροπολογίες και ελάχιστες από αυτές ελήφθησαν σοβαρά από το Συμβούλιο. Τότε βέβαια δεν ίσχυε η συνθήκη της Λισαβόνας. Και το Συμβούλιο τότε, δεδομένου ότι δεν είχαμε τη Λισαβόνα, δεν ενδιαφερόταν καθόλου στο να έχει καλές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή με το Εθνικά Κοινοβούλιο. Στις 17 Ιανουαρίου του 2008 λοιπόν, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που δημιουργούσε την Ευρωπόλ. Αυτή που έχουμε. Αλλά βέβαια η παιδεμή του σώματος ε, εκ μέρους του, του Συμβουλίου δεν σταμάτησαν εδώ. Το περίφημο πακέτο Ευρωπόλ που θα ανέπτυσε την απόφαση του Συμβουλίου Είχε, γιατί τώρα δεν έχει, τέσσερις εισηγητές. Την κυρία Ιντβελτ που θα εξέταζε τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, την ανταλλαγή διαπροσωπικών στοιχείων και την ταξινομημένη πληροφόρηση. Ο κύριος Όλμπριτς, Γερμανός, ήταν εισηγητής για τις τρίτες χώρες και για τους οργανισμούς με τους οποίους θα έπρεπε να συνάψει η Ευρωπόλ συμφωνίες. Ο κύριος Πίρκοφ, ο πρώην υπουργό των Βρετανών Συντηρητικών, εξέτασε το θέμα της μυστικότητας της πληροφορίας. Και εγώ ήμουν εισηγητής για τα δελτία αναλύσεων. Τι συνέβη λοιπόν. Το Συμβούλιο θέλησε να προωθήσει αυτά, αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας που μας έδινε και τις ε, σχετικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό το οποίο δεν θα το ξεχάσει το Κοινοβούλιο. Βέβαια δεν έχει σχέση με την Ευρωπόλ. Εμείς φυσικά και υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Αστυνομία. η οποία δεν έχει σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Χαιρετίζουμε λοιπόν με ιδιαίτερη συμπάθεια όλες αυτές τις πρωτοβουλίες της κυρίας Μάλστρομ, της Επιτρόπου, να εναρμονίσει τα, λεγμένα με τα πεπραγμένα. Όπως είπε και ο Διευθυντής, εμείς εργαζόμαστε με την αξιολόγηση που θα προκύψει μέσα από το νέο κανονισμό, όπως ορίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Όμως πάλι θα πρέπει εδώ να επιστήσουμε την προσοχή σας στην απουσία του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε την τελευταία φορά λέγοντας ότι έξι μήνες μετά από τη θέση σε ισχύ της απόφασης του Συμβουλίου θα έπρεπε να έχουμε την έκθεση, τον απολογισμό και την εφαρμογή, για την εφαρμογή του κανονισμού. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα λειτουργήσει το 2013. Εμείς πρέπει να ολοκληρώνουμε τη διαδικασία αξιολόγησης μέσα από αυτή την πολύτιμη συνεργασία με με τα εθνικά κοινοβούλια για να ολοκληρώνουμε Γι' αυτό λοιπόν τούτων προλεχθέντων το κοινοβούλιο χωρίς να ξεχνάει όλες τις μιζέριες που πέρασε θα πρέπει να προωθήσει τη διαθεσμική συνεργασία. Κατά τη γνώμη μου, ποια θα είναι η κλίδα, ο μοχλός για τη λειτουργία αυτού του κανονισμού. Θα σας αναφέρω τα δύο σημεία τα οποία θα πρέπει αποφασιστικά και θαραλέα να αντιμετωπίζει ο κανονισμός. Το ένα είναι αυτό το οποίο μας μαζεύει εδώ σήμερα, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος είναι ανεπαρκής και ευκαιριακός. Εξαρτάται από το Συμβούλιο βέβαια αυτό. Και δεύτερο, ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο Συμβούλιο έχουμε τον υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε την Εθνική Αρχή Ελέγχου. Και έχουμε την αρχή που θα ελέγχει τον έλεγχο. Όλοι όμως διορισμένοι από κάποιον, διορισμένοι από το Συμβούλιο. Πού είναι λοιπόν η ανεξαρτησία όλων αυτών των οργανισμών, αυτό πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Πρέπει να αποφύγουμε ζητήματα τα οποία θα σας αναφέρω και που εκμηδενίζουν τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εθνικού Κοινοβουλίου. Αυτά τα οποία λέω εγώ λοιπόν δεν έχουν καμία σχέση με όλη αυτή την υποχρεωτική μυστικότητα που απαιτούν τέτοιου είδου εργασίες και που αφορούν στην ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών στη δέκατη, παράγραφο του άρθρου 37. Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό, το πρόγραμμα εργασίας, γενική έκθεση για τις δραστηριότητες σε Ευρωπόλ και μετά λέει αυτά τα έγγραφα θα κατατίθενται στο Συμβούλιο για την έγκρισή τους και το Συμβούλιο θα τα στέλνει αυτά τα έγγραφα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς πληροφόρηση. Ε, πού είναι λοιπόν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η πληροφόρηση δεν είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, 34 παράγραφος 6, ακόμη πιο σοβαρό. Κοινή αρχή θα επεξεργάζεται την έκθεση δραστηριοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα Αυτές οι εκθέσεις θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει σχόλια και τα οποία θα ε, προστίθενται στην έκθεση. Και ακούστε τώρα το φοβερό. Θα αποφασίζει ε, αν θα δημοσιεύει ή όχι την έκθεση δραστηριοτήτων και επιτρέπει τη δημοσίευση κλπ. Μα πού είναι ο έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εσείς κύριε Διευθυντά όλη την υποστήριξη της ομάδας μου την έχετε και όλων μας την έχετε. Εκτιμάμε ιδιαίτερα την εργασία σας. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη, απαράβατη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, παιδοφιλίας, των, της διακίνησης ναρκωτικών, τέλος πάντων. Αυτό ούτε καν το συζητάμε. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να καταγγείλω εδώ και με σκοπό τη συμφιλίωση είναι η ανάγκη το Συμβούλιο να αρχίσει να παίρνει στα σοβαρά το Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ντιέζ Δεμέρα. Και από την Βουλή των Λόρδων τώρα έχουμε τον τρίτο εκπρόσωπο. Θέλω να υπενθυμίσω αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με τις υπηρεσίες διερμηνίας που θα είναι στη διάθεσή μας μέχρι τις 6.30. Αν θέλουμε να συζητήσουμε λοιπόν θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε το πολύ στα 10 λεπτά. Πρόεδρε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που καλέσατε τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να συμμετάσχουν στη συζήτηση με τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή αυτό το απόγευμα και ευχαριστώ που με προσκαλέσετε να μιλήσω για αυτό το θέμα. Η Βουλή των Λόρδων η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που έχουμε στη Βουλή των Λόρδων έχει, λάβει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπόλ πρόσφατα. Επτά εκθέσεις σε 15 χρόνια συνέταξε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε εμπλακεί και παρακολουθήσαμε το έργο της Ευρωπόλ. Και γι' αυτό λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Η τελευταία εκθεσή που δημοσιεύθηκε από την Βουλή των Λόρδων, την Επιτροπή μας στη Βουλή των Λόρδων ήταν το 2008. Μετά από την απόφαση της ε, σύστασης ε, της ε, Ευρωπόλ, της ανασύστασης Ευρωπόλ πριν από την έναρξη σε ισχύ όμως της συνθήκης Λισαβόνας. Ήδη τότε, ήδη στο παρελθόν συνιστούσαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία της Ευρωπόλ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πράγματι και προς τα Εθνικά Κοινοβούλια ακόμα επιπλέον. Και γι' αυτό φυσικά καλωσορίζουμε σε μεγάλο βαθμό κιόλας την επίσημη νομική βάση για την λογοδοσία από πλευρά Ευρωπόλ κοινοβουλευτικά. Και αυτό είναι κάτι πολύ ευπρόσδεκτο. Αυτό το οποίο δεν είναι όμω ευπρόσδεκτο, Πρόεδρε, και πραγματικά τονίζεται στη δική σα εισαγωγή, στη δική σας, από την δική σα κοινοβουλευτική επιτροπή σήμερα το απόγευμα, όταν είπατε ότι είναι θλιβερό ότι ένα έτο μετά από την έναρξη σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, το πλαίσιο αυτό σε σχέση με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί. Το υποστηρίζουμε πλήρω αυτό που είπατε. Και θα ήθελα να επικεντρώσω τι παρατηρήσει μου στο θέμα ακριβώ του κοινοβουλευτικού ελέγχου όχι στις λειτουργίες της Ευρωπόλ και κάποια ευρύτερα θέματα Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορούν θεμητά και νομιμοποιημένα να θυγούν και να καλυφθούν και θα θέλαμε να ζητήσουμε την υποστήριξη της Ευρωβουλής θίγοντας αυτά τα θέματα και συζητώντας τα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από πλευράς μας. Φυσικά δεν είμαστε σε θέση με κανένα τρόπο να κάνουμε τίποτα άλλο παρά αμφισβητούμε την σημασία της διαφορετικής διατύπωσης στο άρθρο 88 που αφορά την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ και του άρθρου 85 όσον αφορά την Eurojust. Και δεν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικές αυτές οι διαφορές, όμως πιστεύουμε ότι διαδικασίες και διεργασίες για την εποπτεία των δύο αυτών οργάνων θα πρέπει να είναι όμοιες και ενιαίες. Θα είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικά χρονοπλαίσια θα έχει θεσπίσει, θα θεσπίζει όσον αφορά την κοινοβουλευτική εποπτεία και έλεγχο των θεσπικών αυτών οργάνων. Πρόεδρε, τον Ιούλιο είχαν προαναγγελθεί τα εξή ε, χρονοπλαίσια όσον αφορά την εποπτεία για την Ευρωπόλ και στην ανακοίνωση που θα έπρεπε να εγκριθεί όσον αφορά τη διαβούλευση 2011. Θα αρχίσουν συζητήσεις συζητήσεις το 2012 θα υπάρξει ένα πλαίσιο και το 2013, τρία χρόνια μετά, θα υπάρξει εξέταση της εποπτείας, εποπτικών δράσεων. Και για την Eurojust θα υποβάλει πρόταση του χρόνου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 2012 θα αρχίσει το πλαίσιο το εποπτικό. Θα ήθελα να ξέρω γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές για τις διεργασίες μεταξύ των δύο και γιατί πρέπει να περιμένουμε για την Ευρωπόλ μέχρι το 2013 για να λειτουργήσει λειτουργήσει αυτή η εποπτεία. Η ΚΟΖΑΚ τόνισε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλεύεται πλήρω με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο. Και εμεί το υιοθετούμε και το υποστηρίζουμε αυτό. Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε ένα απλό πλαίσιο. Οποιαδήποτε διαδικασία και διεργασία θα υιοθετηθεί πρέπει να είναι απλή και πρέπει να είναι ομοιογενής. Τώρα, σε σχέση με την ε, Επιτροπή, δεν έχει την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει υποβληθεί κάποια πρόταση. Αναμένουμε να δούμε ποια πρόταση θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα την εξετάσουμε μέσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού μας ελέγχου και θα την παρακολουθήσουμε και με μια έκθεση που θα συντάξουμε από πλευρά μας. Όμως οι διαδικασίες πρέπει να είναι απλές θα έλεγα. Και όπως τονίζει η Βουλή των Κοινοτήτων, αν σε σχέση με κάθε σώμα ε, κοινοβουλευτικό όταν θα εκπροσωπούνται ε, όταν θα εκπροσωπείται κάθε κοινοβουλευτικό σώμα θα υπήρχαν πάνω από 100 μέλη τα οποία θα συμμετείχαν. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό πιστεύω εγώ. Η εποπτική δομή ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον περίπλοκο χαρακτήρα ε, όσον αφορά και τις δικές μας δραστηριότητες και θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. Δεν είναι δυνατόν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η εποπτεία να δυσχεραίνει το έργο ακόμα περισσότερο. Δεν θέλουμε μια καλή ιδέα να ενταφιαστεί σε γραφειοκρατική επιβάρηση και βάρος. Δεν θέλουμε ο κοινοβουλευτικός ε, έλεγχος ε, να καταλήγει σε εποπτεία αν θέλετε μόνο ατομικού χαρακτήρα θα πρέπει να υπάρχει ενιαία ε, διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, να υπάρχει δυνατότητα βελτίωση ε, των διαδικασιών και να διασφαλίσουμε θα αξίζει τον κόπο το όλο αυτό εγχείρημα. Value for money. Θα πρέπει να είναι σε απλά πλαίσια, να είναι απλή, εξαπλουστευμένη διαδικασία, να μπορεί να λειτουργήσει ταχαίω και εκείνοι που είμαστε υπέρ τη συνθήκη Λισαβόνα και υποστηρίξαμε αυτό το, αυτή τη δράση δίνοντα ε, επιπλέον αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια απογοητεύονται φυσικά όταν τέτοιου είδους χρονοδιαγράμματα προτείνονται για την Ευρωπόλ όπως αυτό το οποίο προτάθηκε. Πρέπει να επανορθωθεί αυτό και να προσαρμοστεί στα σωστά απλά πλαίσια και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία και με τις προτάσεις των βουλευτών. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας βοηθήσατε και με τον χρόνο που πιέζει. Έχουμε ένα σύντομο κατάλογο μελών που θέλουν να παρέμβουν. Έχουμε έξι, θα πάρουμε έναν έβδομο ακόμα. Και αν περιοριστούμε σε... Ναι και εσείς κυρία Ματιέ, εντάξει. Και αν περιοριστούμε το πολύ σε δύο λεπτά ο κάθε αγορητής θα, θα επαρκέσει ο χρόνος και σε σχέση με κάποιες ε, τοποθετήσεις ε, θα, ε, όσων συμμετέχουν στην Προεδρία θα κλείσει μετά η συνεδρίαση. Ο κύριος Σέντσεκ από την Γερουσία της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο και που με προσκαλέσατε επίσης να συμμετάσχω σε αυτές τις διαβουλεύσεις για ε, τα θέματα ε, που αφορούν ε, την Eurojust και τα θέματα δικαιοσύνης. Πρέπει να συζητηθούν αυτά, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να συζητώνται και στα Εθνικά Κοινοβούλια, σίγουρα. Η τελευταία συνθήκη συμπεριλάμβανε αυτό ακριβώς το ζήτημα και μάλιστα σε ένα ε, συγκεκριμένο πλαίσιο και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, ευαίσθητο πεδίο και θέμα για τους πολίτες μας. Πρέπει να είναι λοιπόν ε, εδώ πίσω που βρισκόμαστε εμείς ε, έχουμε πολλούς εθνικούς ε, βουλευτές που συμμετέχουν και αυτό μας ε, πρέπει να ικανοποιεί. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί σε συνάντηση της Κόζακα στο Παρίσι ήδη τον Νοέμβριο του 2008. Μετά στη συνέχεια συζητήθηκε στην Πράγα τον Μάιο πέρυσι. Και αυτές οι, συζητήσεις, ε, αυτές οι συναντήσεις τι κατέδειξαν. Κατέδειξαν ότι η πρακτική εφαρμογή των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων και η λειτουργία τους δεν είχαν επαρκώς αναπτυχθεί. Τώρα όμως κάναμε ένα βήμα παραπέρα και έχουμε προχωρήσει πιο πέρα. Είναι αναγκαίο να ξεκινήσουν τώρα αυτές οι συζητήσεις και να προχωρήσουν όχι μόνο στο επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων αλλά και στο επίπεδο της διακοινοβουλευτικής πλατφόρμας όπως είναι αυτή εδώ η δική μας η διακοινοβουλευτική πλατφόρμα τους επόμενους μήνες πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια ανακοίνωση για τον ε, δημοκρατικό έλεγχο και την λογοδοσία όσον αφορά την ε, Europol θα ήθελα να τονίσω και να αναφέρω τι θα θέλαμε εμείς να γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να βασίζονται στις εκθέσεις της Europol και της Eurojust που ετήσια δημοσιεύονται και που θα πρέπει να είναι διαθέσιμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εμά. Πρέπει να υπάρχει αρκετό χρόνο και για το Ευρωκοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητώνται αυτά τα θέματα, χρησιμοποιώντα τι σωστέ διαργασίε. Να υπάρχει δυνατότητα να τεθούν ερωτήσει προ την Europol και την Eurojust από του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και να συζητηθούν αυτά τα θέματα με του εθνικού εκπροσώπου και φυσικά να βρισκόμαστε σε στενή επαφή και με τους εκπροσώπους στην Eurojust και ε, Europol. Μια καλή πλατφόρμα για αυτές τις συζητήσεις είναι η πλατφόρμα της Κοζάκα. Στη φθινοπορεινή συνεδρίαση της Κοζάκ θα έχουν ε, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις ε, και να κάνουν τα σχόλιά τους. Σας ευχαριστώ. Από την Ιταλική Γερουσία εσείς παρακολουθείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να εκφράσω ε, την αγανάκτησή μου. Πιστεύω ότι το θα πρέπει τώρα που συζητάμε ένα τόσο σημαντικό θέμα και που έχουν ε, συγκεντρωθεί βουλευτές από τόσο μακριά να μας ακούσετε. Η Europol είναι πολύ σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε κάτι το οποίο τόνισε ο εισηγητής Ντεμέιρα όταν αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναθεωρηθεί η απόφαση του Συμβουλίου του 2009. Διότι μέχρι να ρυθμίσουμε τον τρόπο που θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούμε με δημοκρατικό τρόπο. Δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατικούς ε, ελέγχους ε, που να υπόκεινται που, να διεξάγονται από κάποιον ε, εθνικό ή ευρωπαϊκό φορέα. Χρειαζόμαστε ένα σώμα αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στην Ιταλία που να έχει αποκλειστικά αυτό το σκοπό. Η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που θα είναι χρήσιμα για διεθνεί έρευνε θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικού και προσεκτικού χειρισμού από μία αρχή που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να αναλάβει την ευθύνη του, διότι δεν μπορούμε να έχουμε κάποιον διεθνή ή εθνικό οργανισμό ελέγχου πολιτικής φύσεως που να ασχολείται με θέματα μη πολιτικά. Πιστεύω ότι η Europol θα πρέπει να έχει πιο στενές σχέσεις με την Eurojust αλλά και με τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη και γι' αυτό θα πρέπει να ε, εξετάσουμε και το χρονοδιάγραμμα, ε, να, θα πρέπει να μπορούμε να αποφεληθούμε από τις εμπειρίες όλων των κρατών μελών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο στη διαδικασία αυτή. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τη δομή της βάσης δεδομένων της Europol. Θα πρέπει δηλαδή να είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούμε στην ε, Ιταλία για την ε, μαφία ή θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό σύστημα και τι ε, χρήση γίνεται για να ε, αντιμετωπίσουμε τις ε, τρομοκρατικές οργανώσεις. Είμαι μέλος αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα όσα αντανακλώνται από τους συναδέλφους που αναφέρονται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ενδυνάμει εχθρούς από πλευρά της, Euro, της ε, ε, Frontex είμαστε πολλοί που δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την άποψη διότι συμμεριζόμαστε την άποψη των πολιτών που έχουν δικαίωμα, δικαίωμα στην ελευθερία, την ασφάλεια και στη δικαιοσύνη και τουλάχιστον για μένα προσωπική λαμβάνοντας υπόψη ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς προστατεύει αυτά τα δικαιώματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι δική μας ευθύνη να υποστήριξουμε αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες και να υπάρξει πρόοδος στην συνεργασία, όχι μόνο και στις δράσεις, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός. Και αυτό είναι ευθύνη δική μας ως Κοινοβουλίου να ελέγχουμε αυτή την υπηρεσία διότι μόνο έτσι θα προχωρήσουμε στη δημιουργία αυτού του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνη και ασφάλειας. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό επαναλαμβάνοντας χωρίς ε, κάποιες ε, προκαταλήψεις. Ε, και όταν γίνεται λόγος για υπηρεσίες παρακολούθησης, υπηρεσίες ασφάλειας, όλα αυτά πρέπει όμως να είναι υπέρ της ασφάλειας και, της, και των πολιτών. Και μία ερώτηση προς τον Διευθυντή της Ευρωπόλ. Είναι κάτι το οποίο με ρωτάνε οι πολίτες απλοί πολίτες θέλουν να ξέρουν τι γίνεται σε σχέση με την ε, Ευρωπόλ όταν έρχεται η ώρα να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία σε σχέση για παράδειγμα και με την, ε, της ΕΠΑ σε ε, σχέση με πιθανές τρομοκρατικές πράξεις και απόπειρες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβάρας παρακαλώ από τη Βουλή των Ελλήνων. πρόφερα καλά το όνομά σας κύριε Τζαβάρα, σωστά το πρόφερα. Εγώ να μιλήσω. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω το γεγονός ότι σε αυτή εδώ την αίθουσα και κυρίως στις αίθουσες των Εθνικών Κοινοβουλίων αυτό που αποτελεί ύψιστη υπηρεσία στη δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τη δημοκρατία του καιρού μας, είναι ο σεβασμός και η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί στοιχείο του ιδεολογικού προτάγματος το οποίο όλοι υπηρετούμε, η αναγνώριση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί δε και στοιχείο της ένομης τάξης όλων των κρατών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επομένως δεν μπορώ να κατανοήσω την τάση που έχουν μερικοί συνάδελφοι να μονοπολούν την συνηγορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ που είμαστε σήμερα αυτό που πρέπει να επιβεβαιώσουμε είναι η ικανότητά μας να μπορούμε να γινόμαστε χρήσιμοι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη μια μεριά συγκρούσεις όπου από τη μια μεριά συγκρούονται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη μεριά συγκρούεται η προσπάθεια που κάνουμε όλοι για έναν καλύτερο κόσμο έναν κόσμο ασφάλειας ελευθερίας και δικαιοσύνης επομένως όλες αυτές οι ταυτολογίες που ακούγονται δεν προσφέρουν ούτε και προωθούν το δημοκρατικό διάλογο. αυτό όμως που θα ήθελα να ρωτήσω το διευθυντή της europol που έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα και είναι τιμή μας να τον ακούμε είναι το πώς μέχρι σήμερα και ειδικά για θέματα που έχουν σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων αυτών αλλά κυρίως με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και μάλιστα του εγκλήματος το οποίο έχει ουσιαστικά προαχθεί και υπό την έννοια ότι έχουν καταργηθεί τα εθνικά σύνορα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως έχουν κατά αυτόν τον τρόπο αποδεσμευτεί και τάσεις εγκληματικών οργανώσεων να αναπτύσσουν τέτοιου είδους δραστηριότητες σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Πώς μπορεί αυτή η συνεργασία μεταξύ των κρατών των εθνικών αφενός από την άλλη μεριά της Europol και από την εκτρίτου άλλες οργανώσεις όπως είναι η οργάνωση για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος πώς μπορούν αυτό να συνεπάρξουν και το λέω γιατί έχω στο νου μου το πολύ σοβαρό θέμα που μας απασχολεί στην Ελλάδα για την αποκάλυψη της αλήθειας που έχει με την παράνομη δράση της Siemens στην Ελλάδα όπου εκεί κατάφερε από το 1996 αυτή η γερμανική επιχείρηση να διαφέρει υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πλήγμα και στο δημόσιο χρήμα αλλά κυρίως και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τέτοιων νοουμένων των δικαιωμάτων που έχει ο πολίτης να απαιτεί από την κυβέρνησή του αποτελεσματικότητα και προσπάθεια ανταπόκρισης σε όλα τα αιτήματα που στηρίζονται στον νόμο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσου συμμετείχαν στο πάνελ για τι παρουσιάσει του και για του συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων που δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να τους πω ότι όταν πρόκειται για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς Europol και Eurojust ιδιαίτερα ενώ οι ευρωβουλευτές ήταν υπέρ του να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες σε αυτές τις υπηρεσίες και οργανισμούς και στην Europol το Συμβούλιο ήταν πολύ πιο διστακτικό, ήταν πολύ πιο επιφυλακτικό. Και για παράδειγμα ο συνάδελφος Αγουστίν Μέρα έδωσε ένα καλό παράδειγμα για αυτά από πλευράς του. Ερώτησή μου και για τον Διευθυντή της Europol και για τον εισηγητή μας κύριο Ντεμέρα. Η ερώτησή μου είναι πού βρισκόμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εμπιστοσύνη του Συμβουλίου. Και όταν λέω Συμβούλιο, φυσικά εννοώ τα κράτη-μέλη, έτσι. Αυτό είναι. Τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Τι γίνεται από πλευρά τους με την εμπιστοσύνη τους εναντί της Europol. Γιατί υπάρχει αυτή η διστακτικότητα, η επιφυλακτικότητα. Μήπως επειδή δεν θέλουν να δώσουν, να απεμπολίσουν τα δικαιώματα ελέγχου από πλευρά τους στα κράτη-μέλη όσον αφορά παράδειγμα ανακριτικές δραστηριότητες ή ερευνητικές δραστηριότητες ή δεν έχουν εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς. Φυσικά εκείνοι που είναι υπεύθυνοι είναι υπεύθυνοι ε, υπάλληλοι αστυνομικών ε, οργάνων των κρατών μελών. Αν κάτι τέτοιο λοιπόν συμβαίνει, τότε θα πρέπει να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί αυτή η έλλειψη, η απουσία εμπιστοσύνη. Και το ερωτώ αυτό επειδή πρόσφατα τις τελευταίες μέρες ε, στο παρελθόν ήμουνα στην Κολομβία τις προάλλες και όχι μόνο είχαμε υπαλλήλου ε, της ε, κυβέρνηση, αλλά και εκπρόσωποι των think tanks των ε, ομάδων προβληματισμού χαιρέτησαν την εταιρική σχέση συνεργασίας μεταξύ Europol και αρχών της Κολομβίας και φυσικά σίγουρα με πολύ φροντίδα και μέρημνα το έκαναν αυτό από πλευρά τη Europol διότι κανένα δεν διακινδυνεύει τη ζωή των υπαλλήλων του έτσι χωρί ε, λόγο και αξία. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη σε σχέση με την Europol. Ο κύριος Καλασεύσκη, μέλος της ε, Πολωνικής Βουλής παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Για να ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την άποψη του ε, Λόρδου της Βουλής των Λόρδων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε οι διαδικασίες, οι διεργασίες για τη Eurojust και τη Europol με την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας να είναι διαφορετικές οι διεργασίες για τη Europol και για την Eurojust. Διαφορετικές και με διαφορετικά χρονοπλαίσια και ειδικά είπε ο εκπρόσωπος, ο διευθυντής της Europol ότι σε σχέση με την δυνατότητα προσαρμογής των ε, λειτουργιών της ε, Europol ε, που μέσα σε αυτό το πλαίσιο τίθεται θα ήθελα να επανέλθω σε κάτι εγώ και να αναφέρω ότι κάποιοι από τους προλαλήσαντες είπαν ότι η συλλογή η συλλογή των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να είναι μέρος, μήμα των εργασιών και δράσεων της Frontex. Εγώ είμαι εναντίον μιας τέτοια πρότασης, διότι η συλλογή και αποθήκευση, η συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο. Θα μπορεί να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα και στοιχεία η Frontex, αλλά δεν θα πρέπει να μπορεί να τα συλλέγει ή η ίδια να μπορεί να τα αποθηκεύει από πλευρά τη. Έχω όμω ε, μία ερώτηση προ τον διευθυντή τη Europol. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη συνεργασία μεταξύ Europol και Frontex. Ιδιαίτερα όσον αφορά διασυνοριακέ, διαμεθοριακέ ε, δράσει καταπολέμηση εγκλήματο. Για παράδειγμα, καταπολέμηση ε, λαθρεμπορίου ανθρώπων, ναρκωτικών κτλ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Μούλντε, παρακαλώ, τη Επιτροπή Λίμπε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Έχω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Στην συνθήκη της Λισαβόνας γίνεται λόγος για έναν Ευρωπαίο εισαγγελέα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, παράσιτα από κινητό τηλέφωνο. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τη δουλειά της Europol αν υπήρχε ένας τέτοιος θεσμός τι θα γινόταν τελικά και τέλος η κυρία Ματιέ της Επιτροπής Λίμπε παρακαλώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα τη γνώμη του Διευθυντή της Europol για τη ΣΕΠΟΛ Ξέρετε ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ε, απέρριψε την απαλλαγή του προϋπολογισμού για τη ΣΕΠΟΛ του 2008 Λοιπόν υπήρξε ομοφωνία στην απόρριψη της απαλλαγής και θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται ο διευθυντής της Europol για αυτό το σπάσιμο σταδίο της κατάρτισης των αστυνομικών. Δεν θα έπρεπε η Ευρωπόλ να είναι αρμόδια γι' αυτό. Ήδη δημιουργεί ένα πρόβλημα η έδρα της ΣΕΠΟΛ για το προσωπικό κτλ. Αφήστε δε που είναι και μόνο τρία μέλη, τρει, τρεις υπάλληλοι ΣΕΠΟΛ. Οπότε φαντάζομαι και λόγω μεγέθους ε, δεν είναι αποτελεσματική η κατάρτιση των αστυνομικών. Δεν θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να συγκεντρωθούν στην Ευρωπόλ. Φυσικά με όλα τα μέσα ad hoc ε, που χρειάζεται ο οργανισμός σας ε, για να τα διευθύνει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχουν πάλι οι ομιλητέ μας, οι συγκητέ μα. Ε, θα ήθελα όμω, λέει ο πρόεδρο εκ των προτέρων, να ευχαριστήσω του ε, διερμηνεί που θα μα χαρίσουν μερικά επιπλέον λεπτά ώστε να προλάβουμε. Παρά την πίεση χρόνου. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, και δίνω πρώτα το λόγο στον Διευθυντή της Europol, τον κύριο Wainwright. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να καλύψω όσο γίνεται περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Κάποιες παρατηρήσεις έγιναν σχετικά με την αξιοπιστία της Europol. Η κυρία Weber ε, το ανέφερε αυτό ε, καθώς και άλλοι. Είναι αλήθεια ότι μετά από 15 χρόνια προσεκτικής ανάπτυξη, η Europol πρέπει ακόμα να ε, παλεύει για τη θέση της ε, για να ε, χαίρει εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Φυσικά τα πράγματα είναι καλύτερα, φυσικά συνεχίζουν να βελτιώνονται τα πράγματα. Η ο παρόν ρυθμός εργασία μας, 15.000 ε, υποθέσεις το χρόνο, είναι ε, σαφώ αυξημένο σε σχέση με πέρσι, αλλά ε, ιδιαίτερα στον τομέα της τρομοκρατία υπάρχει ακόμα επιφύλαξη από τις εθνικές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες της Europol στον τομέα αυτών. Γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ ευαίσθητο ε, τομέα εργασίας. Ε, έχουμε να κάνουμε με τρομοκρατία, έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητε πηγέ πληροφοριών, έχουμε να κάνουμε με μια κοινότητα που είχε πολλές επιτυχίες ε, τα τελευταία χρόνια. Η η πρόοδος στην Ευρώπη έχει σημειωθεί σε διμέρες επίπεδο. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί η Europol αρκετά και γι' αυτό υπάρχει εδώ ένα εμπόδιο που έχει να κάνει με την οτροπία που θα πρέπει να ξεπεραστεί. Ε, η εικόνα του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σίγουρα αλλάζει, γίνεται πιο παγκόσμια, πιο το επιχείρημα λοιπόν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά ε, όργανα όπως η Europol ε, γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Θα πρέπει να πετύχουμε την εμπιστοσύνη των ε, συναδέλφων μας ε, για να ε, πετύχουμε την προστιθέμενη αξία. Η βάση δεδομένων, για παράδειγμα, της Europol είναι μοναδική στην Ευρώπη. Μόνο η Europol έχει τέτοια επισκόπηση των πληροφοριών για τις ε, εγκληματικές δραστηριότητες και τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Ευρώπη στο σύνολό της. Έχουμε λογισμικό υψηλής τεχνολογίας και γενικά εξοπλισμό που μας βοηθάει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο επικίνδυνα ε, εγκληματικά και τρομοκρατικά δίκτυα. Κάθε φορά που έχουμε κάποια μεγάλη επιτυχία, πετυχαίνουμε λίγο, λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη από τους συναδέλφους μας που κάνουν έρευνα. Πιστεύω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να μας βοηθήσει, διότι έχει να κάνει και με τους εθνικούς νομοθέτες, τις αρχές σε εθνικό επίπεδο, διότι οργανισμοί όπως η Europol θα πρέπει να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Και να απαντήσω σε μια άλλη συγκεκριμένη ερώτηση. Η σχέση μας με τη Frontex ήδη είναι πολύ ισχυρή. Ε, νομίζω ότι ο κ. Λάτινεν ήδη το είπε αυτό. Η ικανότητα της Europol να χρησιμοποιεί ε, τις δυνατότητες της ε, για ε, κεντρική πληροφόρηση, να παρέχει αναλύσεις ώστε να γίνεται σωστή κινητοποίηση ε, των, ε, των δυνάμεων και σε κάποιους συγκεκριμένους ε, τομείς η Europol και η Frontex συνεργάζονται πολύ στενά. Ο κύριος Μάλτερ ρώτησε σχετικά με τον Ευρωπαίο εισηγητή. Έχουμε μια πολύ επικοτομητική συνεργασία με την Eurojust ήδη. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και η δουλειά η δική μας συμπληρώνεται πολύ καλά από τη δυνατότητα της Eurojust να ολοκληρώσει την, ε, την κάθε υπόθεση με τη δικαστική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή Ευρωπα... Ευρωπαίο εισαγγελέα, αλλά δεν το αποφασίζω εγώ. Εάν ε, το έχουμε τελικά, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πλαισιώσουμε το ρόλο του και σε αστυνομικό επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή να τεθεί το ερώτημα κατά πόσο θα συμπληρωθεί η εικόνα των ε, νομικών ε, αρμοδιοτήτων της ε, Europol. Επίσης, όσον αφορά τη ΣΥΠΟΛ, συμφωνώ ότι η ΣΥΠΟΛ βρίσκεται υπό πίεση και η αδυναμία της, του Κοινοβουλίου να χορηγήσει απαλλαγή δείχνει ακριβώς αυτό. Όπως και η δική μου υπηρεσία, η ΣΥΠΟΛ χρειάζεται έναν σωστό κανονισμό προσωπικού και δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι όμω πολύ δύσκολο το έργο με του ε, πολύ περιορισμένου πόρου που έχει. Τη βοηθάμε όσο μπορούμε, ε, εκμεταλλευόμενοι τι ε, συνέργειε τη ΣΥΠΟΛ με τη Europol. Ε, μόλις συμφωνήσαμε με τον νέο ε, διευθυντή, τον κύριο Μπάνφη, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα. Και ε, είπαμε ότι θα κανονίσουμε μια μεγάλη αστυνομική διάσκεψη στα ε, γραφεία της Europol. Κάνω λοιπόν ό,τι μπορώ για να εκμεταλλευτώ τις φυσικές συνέργειε που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο υπηρεσίε μας. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι ίσως η πιο σημαντική και έχει να κάνει με ε, αυτό που είπε ο κύριος Τσαβάρας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι μια υπηρεσία σαν την Europol θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και, την, ε, και την ασφάλεια, την ελευθερία και την ασφάλεια. Αυτές είναι ε, αλληλοσυμπληρώμενες έννοιες στην κοινωνία μας και πιστεύω ότι στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε ε, ε, ε, να προστατεύσουμε το βασικότερο ανθρώπινο δικαίωμα όλων μας, το δικαίωμα της ζωής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας με υπεύθυνο τρόπο και πιστεύω ότι ο τρόπος που το κάνουμε θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τους διερμηνείς για το χρόνο που μας δίνουν. Είναι οι καλύτεροι διερμηνείς του κόσμου σε αυτό το κοινοβούλιο, λέει ο κύριος Διεθνεμέρα και οι διερμηνείς αισθάνονται αμήχανοι. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, Κοσάκ και όπως είπε και ο Ιταλός συνάδελφος θα πρέπει να εμβαθύνουμε πάρα πολύ στον δημοκρατικό έλεγχο βελτιώνοντας την απόφαση του Συμβουλίου μέσα από τον κανονισμό Επίσης στον κύριο στον κύριο Τζαβάρα πρέπει να πω ότι όλα αυτά δεν είναι περιουσία κανενός. Εμείς έχουμε σήμερα στο πρωτογενές δίκαιο το, τα, τα, τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης για την εμπιστοσύνη τώρα στα κράτη-μέλη. Μα η εμπιστοσύνη έγκυται ε, στον καταμερισμό πληροφόρησης και δεδομένων. Θα πρέπει εμείς να επεξεργαζόμαστε, να αναλύουμε και να ανταλλάσσουμε δεδομένα. Γι' αυτό μας χρειάζεται επαγγελματισμός και εξειδίκευση. Αυτό έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων υπηρεσιών των κρατών μελών και μετά εμπιστοσύνη μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωκοινοβουλίου για να μπορέσει η Ευρωπόλ να έχει μεγαλύτερη νομιμότητα και θα πρέπει να θεωρείται κάτι το απόλυτα αυτονόητο ο δημοκρατικός έλεγχος χωρίς επιφυλάξεις. Εμείς θα σεβαστούμε και τις εργασίες και τη μυστικότητα της Ευρωπόλ. Και κάτι άλλο σχετικά με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ο συνάδελφος που ανησυχεί για αυτό το θέμα. Εγώ του εύχομαι ένα βέβαιο ε, μέλλον ε, από χωροχρονικής πλευράς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ελπίζω θα με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι αν θα είμαι πολύ σύντομος και περιορίσω τα σχόλιά μου στο θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου θεωρώ εγώ με σεβασμό σε όλα τα σημαντικά θέματα και παρατηρήσεις που έγιναν ότι αν ακολουθήσουμε όλες τις παρατηρήσεις και σχόλια σε όλη αυτή την ευρύτερη συζήτηση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο θα πάμε ακόμα πιο πέρα και πιο μακριά από ότι ήδη σήμερα βρισκόμαστε που είμαστε πολύ μακριά ήδη. Και εμείς που είμαστε υπέρ της ε, Europol ελπίζω ότι η αμοιβή εμπιστοσύνη θα αυξηθεί και σίγουρα όλοι οι εκπρόσωποι στην Europol θα πρέπει να έχουν ε, ας το πω έτσι, έγκριση από πλευράς ε, ε, ασφαλείας για να μπορούν να ικανοποιηθούν και να καθησυχάσουν τα κράτη-μέλη. Αλλά επανέρχομαι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εξετάζουμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να δουν τα θέματα στρατηγικής και θα μπορεί να υπάρχει αποτελεσματικότητα, value for money. Κάνουμε λόγο για λογοδοσία και πρέπει να ξεχωρίζουμε τα θέματα λογοδοσίας από τα θέματα ελέγχου, αυστηρά θέματα ελέγχου αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ όλους αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη. 3,5 ώρες ε, έντονη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακόμα μας περιμένουν από αύριο από τις 9 στις 12.30 άλλες 3,5 ώρες. Προσβλέπουμε στην δεύτερη αυτή συνεδρίαση για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και ας κλείσω αυτή τη πρώτη συνεδρίαση εργασίας ευχαριστώντας τους διερμηνείς και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει δεξίωση με ποτό κόκτέιλ. Σας προσκαλώ όλους σας, ευρωβουλευτές, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων εκπροσώπους, κάτω θα έχουμε στο δεύτερο όροφο δεξίωση που θα ξεκινήσει τώρα και σας ευχαριστώ όλους σας.